Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Κύριε Κλίντς, μπορούμε να συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λείπει ο Πρόεδρος, λείπουν οι Αντιπρόεδροι έχει φτάσει και η δική μου σειρά να αναλάβω την Προεδρία της Επιτροπής μας. Θα ξαναξεκινήσουμε τώρα. Συνεχίζουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Εδώ θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μοργάνο Λουίτζι. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί. Γιατί επιθυμούμε να δούμε τι έχει πει και η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Έχετε το λόγο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες και για τη δουλειά που έχουν κάνει και για το υλικό το οποίο μου έχουν καταθέσει. Έχουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις που λάβαμε και έχουμε επίσης και κάποια διορθωτικά σχόλια. Θέλω να κατανοήσετε πως οι ίδιοι πόροι είναι όχι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και πολιτικό. Δηλαδή, θέλουμε ή όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα απαραίτητα μέσα για να μπορεί να εξυπηρετήσει τις φιλοδοξίες της. Είμαστε Ευρωπαίοι και πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον μας και στο άμεσο μέλλον και στο ε, μακροπρόθεσμο μέλλον. Τι επιθυμούμε να γίνει και θα πρέπει να ε, αντιδράσουμε ε, σε αυτή την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι δική μας η απόφαση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που επηρεάζουν το μέλλον της Ευρώπης. Και εγώ ως εισηγητής και οι προσπαθήσαμε οι τροπολογίες ε, που θα εντάξουμε στο κείμενο να αποδεικνύουν πως θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να μοιραστούμε ε, χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε η προσέγγιση την οποία προτείνω εγώ και την οποία νομίζω συμμερίζονται και οι υπόλοιποι σκιώδεις εισηγητές είναι όχι μόνο να πούμε ποιοι πόροι μας φαίνονται ότι αποτελούν προτεραιότητα, αλλά να εξηγήσουμε και για ποιο λόγο αυτοί η οι πόροι είναι προτεραιότητα και πώς θα χρησιμοποιηθούν και θα τους διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω πως κάποιοι συνάδελφοι είναι κατά της προόδου προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα συνέστημα το οποίο εγώ δεν συμμερίζομαι και θεωρώ πως είναι και επιβλαβές για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά το σέβομαι και όποτε χρειάζεται είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Τώρα υπάρχει κάτι το οποίο με έχει εκπλήξει. Δηλαδή, το ότι είχαμε αρκετές δυσκολίες στη στιγμή της διαπραγμάτευσης με κάποιες ομάδες οι οποίες παρόλο που είναι υπέρ και παρόλο που έχουν τις ευρωπαϊκές και παρόλο που έχουν συνεισφέρει στην κατασκευή αυτής παρόλα αυτά δεν θέλουν το κοινοβούλιο να έχει πιο δραστήριο ρόλο στο χώρο αυτό. Πάρα πολύ περίεργο αυτό γιατί εμείς εκπροσωπούμε εδώ τον Ευρωπαίο πολίτη. Βεβαίως κατανοώ πως τελικά χάρη στη δουλειά που έχουμε κάνει όλοι μας, καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Και μπορεί βέβαια να μην είναι τόσο φιλόδοξο το κείμενο όσο θα ήθελα εγώ, αλλά βάζουμε ένα ξεκάθαρο στόχο προς τον οποίο θα κινηθούμε ε, στο μέλλον ε, με τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό έχει λάβει υπόψη όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε στους ίδιους πόρους και νομίζω ότι καλύπτει τα σημεία τα οποία είναι ευαίσθητα για τις περισσότερες ομάδες. Γι' αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους για ό,τι έχουν κάνει και είμαι στη διάθεσή σας να συνεχίσουμε, να συνεργαζόμαστε και θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και ελπίζω πως η ψηφοφορία αργότερα θα πάει καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάλη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να σας πω πως είμαστε ικανοποιημένοι που φτάσαμε ε, στους συμβιβασμούς αυτούς ε, μέσα στην έκθεση, οι οποίοι βεβαίως δεν μας ικανοποιούν πλήρως. Όλοι χρειάστηκε να δεχτούμε σημεία ε, συμβιβαστικά, αλλά τελικά Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα κοινό παρανομαστή κατανόησης για το ποια θα πρέπει να είναι η θέση μας σχετικά με το θέμα των, ε, του συστήματος ίδιων πόρων. Ε, έχουμε δύο μεγάλα κενά που θα χρειαστεί να καλέψουμε στον προϋπολογισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Το ένα είναι τα νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες και το άλλο είναι το Brexit. Οπότε για το λόγο αυτό έγινε και αυτή η πολύ έντονη συζήτηση για το νέο σύστημα. Όλοι θέλαμε στη γνωμοδότηση να φαίνεται πως η μεταρρύθμιση του συστήματος για τους ίδιους πόρους δεν θα πρέπει να επιβάλλουν ένα νέο φορολογικό βάρος στους πολίτες μας και ότι θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα σταδιακής ε, κλιμάκωσης των, του συστήματος, το οποίο θα παραδίδει ε, πλεονεκτήματα για όλους τους πολίτες στα πλαίσια ε, του πλαισίου, στα πλαίσια του συστήματος που έχουμε, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τους επανυπολογισμούς, επανυπολογισμούς που θα γίνουν για κάποια χρηματοδοτικά, ε, χρηματοδοτικές εκκρεμότητες και βέβαια με απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες. Έχουμε κάποιες γραμμές στον υπολογισμό που θέλουμε εμείς να στηρίξουμε και για τις οποίες έκανα εγώ συζήτηση με τον Επίτροπο κύριο Έτιγκερ και να σας πω πως και αυτός μου τόνισε πως η άποψη του ταυτίζεται με τη δική μας. Δηλαδή, θα πρέπει να παραμείνει ενιαίος ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και δεν χρειάζεται δεύτερος επιπλέον προϋπολογισμός. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ε, ενιαίο προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες και των 27 κρατών μελών. Αυτή είναι η θέση μας, αυτό πρέπει να τονίσουμε και νομίζω ότι η συγγνωμοδότηση αυτό φαίνεται. Επίσης, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να είναι πιο αποδοτικές οι δαπάνες μας. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε να υπάρχει ε, σαφής ε, συσχετισμός μεταξύ δαπάνης και ε, ευκταίου στόχου και νομίζω ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη παράλληλα με την προσπάθεια που θα κάνουμε για ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Σε επόμενες συζητήσεις που θα γίνουν στο Κοινοβούλιο θα δείτε πως θα εξαρτηθεί και από τις άλλες επιτροπές το πώς θα καταλήξει το θέμα αυτό και αν έχουμε νέες πηγές εσόδων. Πάντως η θέση μας εδώ είναι πολύ σαφής και ελπίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τη λάβει δεόντως υπόψη της. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για αυτή την πρόταση και για τη στάση του στο πλαίσιο των πρώτων συνεδριάσεων ε, με τους κοιόδης συζητητές ε, καθώς ήταν πολύ συνεδριάσιμος. Κατά τη δική μου άποψη δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε μια φάση όπου η έκθεσή μας ανταποκρίνεται ε, στα όσα θέλει να εκφράσει η Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, και αυτό γιατί σε μεγάλο βαθμό έκθεση δεν εστιάζει στο πραγματικό θέμα της. Ε, με τον τρόπο δηλαδή που έχει συνταχθεί αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί μια έκθεση σε σχέση με τους ίδιους πόρου τα έσοδα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια έκθεση αντιθέτω ε, που εστιάζει κυρίως στις δαπάνες ε, της Ένωσης, δηλαδή νέα σχέδια, νέα project τα οποία θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε, το την προπολογισμό τη Ευρωζώνη και ούτω καθεξή. Ουσιαστικά δηλαδή εστιάζει πολύ στι δαπάνε και όχι στου ίδιου πόρου που αποτελεί βέβαια το αντικείμενο εξέταση ε, τη Επιτροπή μα. Από εκεί και μετά υπάρχουν μια σειρά από παρατηρήσει που γίνονται σε ό,τι αφορά τι ε, καινοτομίε, θεσμικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε έναν Υπουργό Οικονομικών ή όχι, όλα αυτά δεν σχετίζονται με το ζήτημα των ιδιών πόρων της Ένωσης. Κατά δική μου άποψη, ε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για τις δαπάνες της Ένωσης. Ε, γιατί δεν θα πρέπει να αναφερθούμε μόνο ε, στις ε, νέες ε, αρμοδιότητες που καλείται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και υφιστάμενες αρμοδιότητες οι οποίες διευρύνονται σε κάποιο βαθμό. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε τώρα να παρατηρεί η Γαλλία σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική. Όλα όμως αυτά δεν αποτελούν αρμοδιότητες της δικής μας Επιτροπής, κατά συνέπεια δεν καλούμαστε εμείς να τοποθετηθούμε από αυτόν. Ποιο είναι το ζητούμενο για μας, με ποιο ζήτημα θα πρέπει να ασχοληθούμε και το οποίο δεν θίγεται στην έκθεση είναι το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρο τη από ιδίου πόρου ακριβώ, από την επιβολή δηλαδή φόρων από την ίδια την Ένωση, ή εάν θα πρέπει η χρηματοδότηση τη Ένωση να συνεχίζει να ε, υποστηρίζεται και από του υπολογισμού των κρατών μενών με βάση δηλαδή το ποσοστό του ακαθάριστου του εθνικού εισοδήματό του. Ε, άρα λοιπόν αυτό το σημαντικό ζήτημα δεν συζητάται μέσα στην έκθεση. Ε, και μάλιστα εγώ ε, δεν είμαι ε, πεπισμένος ότι πράγματι αυτή η ενίσχυση του προπολογισμού της Ένωσης από τους εθνικούς προπολογισμούς βάσει του ε, ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος είναι η ενδεδειγμένη λύση. Ουσιαστικά δηλαδή αν συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο δεν ακολουθούμε την σωστή λογική την οποία θα έπρεπε να ακολουθούμε. Βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο είναι αρμόδια ούτω ή άλλω για τη συλλογή των φόρων τα κράτη-μέλη και όχι η Ένωση. Άρα λοιπόν, ω προ αυτό το ζήτημα, η έκθεση δεν θεωρώ πω έχει ε, φτάσει εκεί που θα έπρεπε και ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, υπάρξουν ακόμα σημαντικέ βελτιώσει τη έκθεση, τι οποίε πραγματικά ελπίζω πω θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ. merci. Wolf euh, äh, äh, Έχεις πάρει τη θέση του Ενρίκε. Όχι, δεν αντικαθιστώ κανέναν, δεν είμαι σχεδόν εισηγητή, ούτε μιλώ εκ μέρου του εισηγητή. Για μένα τον ίδιο παίρνω το λόγο. Και θα πρέπει ευθύ εξ αρχή να ομολογήσω ότι δεν έχω εντρυφήσει στο ζήτημα, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει συμπληρωματικά προς τα όσα είπε ο συνάδελφος Λούκα. Έχω την αίσθηση ότι κάνουμε το ίδιο ασφάλμα με αυτό που κάναμε πρόσφατα. Δηλαδή όταν δεν έχουμε τους απαραίτητους ε, πόρους, τα απαραίτητα κονδύλια, δεν διαρωτώμαστε ως προς το πώς μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερη αποδοτικότητα σε ό,τι αφορά την χρήση των υφιστάμενων ε, ε, κονδυλίων, αλλά αντιθέτω εστιάζουμε στο πώς μπορούμε να ε, συλλέξουμε συμπληρωματικά κονδύλια. Άρα λοιπόν θεωρώ πως κάνουμε το ίδιο σφάλμα και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μέσω τροποποιήσεων στο σύστημα του φόρου προστιθέμενης ε, αξίας, μέσω της θέσπισης μιας κοινή ενοποιημένης φορολογικής βάσης εταιριών, να θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα νέα κονδύλια, παρότι η εμπειρία μας δείχνει ότι παρότι έχουμε ασχοληθεί για πολύ καιρό με αυτό το ζήτημα, δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Δηλαδή το να θέσουμε σε διαφορετική βάση την, ε, το φόρο προστέμενας αξίας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της απάτης ΦΠΑ, ε, το οποίο βέβαια μας οδηγεί σε απόλυες, σε διαφυγόντα ε, έσοδα ε, υψηλότατα, είναι κάτι επί το, οποίο, δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε και σε ό,τι αφορά την CCCTB μπορώ να θυμηθώ ότι ο Τσάλι Μαγκρίδη ο οποίος ήταν επίτροπος από το 2004 στο 2009, είχε κάνει τα πάντα ούτως ώστε να επιτύχει την επιβολή αυτής της κοινή βάση, αλλά δεν τα κατάφερε και πιστεύω πως θα επαναληφθεί το ίδιο σενάριο. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να εκχωρήσουν αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τον τομέα ακριβώ το, φορολογικό και ειδικότητα την, την ε, συλλογή των φόρων. Ε, ακόμα δηλαδή και αν ουσιαστικά το δεν ρυθμίζουμε κάτι σε, σε ό,τι αφορά την εθνική νομοθεσία, αλλά μόνο ένα συγκεκριμένο φορολογικό συντελεστή, παρόλα αυτά τα ε, κράτη-μέλη φοβούνται πάρα πολύ ε, ω προ αυτή την παρουσίαση στην αρμοδιότητά του και δεν το επιθυμούν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο προσεκτικά το τι, ε, προσεκτικότερα το τι θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι θεσμικέ μεταρρυθμίσει, δηλαδή το ESM να ε, καταστεί ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αν θέλουμε πράγματι να έχουμε αντί για επίτροπο ένα Υπουργό Οικονομικών τη Ένωση και ούτω καθεξής, όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Και πράγματι με την ανάληψη για παράδειγμα των ε, ζητημάτων των εξωτερικών υποθέσεων από μία είπατε εκπρόσωπο ε, είχαμε ένα, μία επιτυχημένη περίπτωση. Οπότε εάν θα μπορούσαμε να αναθέσουμε και ένα τέτοιο πόστο σε κάποιον τον Υπουργού Οικονομικών πράγματι θα είχε τα πλέον εκτιμάτά του. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτός ο νέος θεσμός δεν θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός ε, προς ε, δηλαδή τον, τον επιτρόπου. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα δημιουργούσε ε, ουσιαστικά μόνο επιπρόσθετες ανάγκες ψηφοφοριών, κατανομής αρμοδιοτήτων και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στείλει κανεί ε, το λόγο από την ΚΟΕ, από του πράσινου. Θέλει κανεί άλλο το λόγο για την έκθεση Μορκάνο. Έχετε το λόγο, κύριε Συνσηγητά. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τις ε, τοποθετήσεις που ξαναδιατυπώνουν τις ίδιες ε, προτάσεις που μας έχουν φέρει στο κείμενο αυτό. Σήμερα πρέπει να πω, σήμερα το πρωί άκουσα ε, τους προσκεκλημένους της Επιτροπής των Προϋπολογισμών, τον Επίτροπο Oettinger βεβαίως που έχει τοποθετηθεί για το θέμα και δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα να εντοπίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις που απασχολούν βέβαια και την Επιτροπή μας συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ε, ιδεών που μου επιτρέπουν να υπενθυμίσω και να τονίσω πάνω απ' όλα το ρόλο της ομάδας υψηλού επίπεδου η οποία εντόπισε συγκεκριμένε ε, προτάσεις σε σχέση με τα όσα έχει πει η Επιτροπή των Προϋπολογισμών και που πρέπει να προσδιορίσουμε για τον φόρο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για ένα τέλος για τη χρήση των πλαστικών, αλλά και γενικότερα μια ιδέα που υποδεικνύει ότι για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και σε σχετικούς αλλά και σε απόλυτους όρους να ενισχύσει την χρηματοδότηση και για το γενικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1 στο 1,1, 1,2, 1,3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λογική λύση γιατί βεβαίως υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων που μπορεί να θεωρούν ότι μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να περιοριστεί σε ένα πλαίσιο για το οποίο γνωρίζουμε ότι ήδη καταγράφονται διαφορετικές ε, προτάσεις και που και εκείνων που λένε ότι το κοινοβούλιο είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει από τις εκθέσεις του να διευκρινίσει και να υποστηρίξει μια πολιτική επιλογή ουσίας. Γιατί είναι δύσκολο να, δούμε, να βρούμε τη χρυσή τιωμή μεταξύ εκείνων που θέλουν να περιορίσουν το ειδικό βάρος της, της Ένωσης σε σχέση με εκείνους που θέλουν ακριβώς το αντίθετο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διότι νομίζω ότι έπρεπε ακριβώς να γίνει αυτή η αντιπαράθεση επί της ουσίας των προτάσεων για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία λοιπόν για τη γνωμοδότηση σε λίγο όταν αρχίσουν οι ψηφοφορίες και περνώ στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση για τα σημεία 8, 9, 10 και 11 της ημερήσιας διάταξης ε, το πρώτο ε, θέμα είναι είναι αυτό το σχετικό με τις ε, εποπτικές αρχές, ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, Τραπεζική Αρχή, στο πλαίσιο της ΜΥΦΙΤ και της ε, ε 2, το τρίτο κείμενο που αφορά την ε, μείωση του συστημικού κινδύνου και την πρόταση για, τον, ε, για την τροποποίηση της έδρας Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ο Μπουρχαρτ Πάλτς συνεισηγητής λαμβάνει το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία συνεισηγητρία και προσωρινή πρόεδρε. Ο συνεισηγητής βεβαίως χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεση αυτήν που έχει να κάνει με την αναθεώρηση των εποπτικών αρχών. Τις τελευταίες εβδομάδες ετοιμάσαμε μας με την σε ένα έγγραφο εργασίας, το διαθέσαμε χθε στα μέλη. Ένα έγγραφο το οποίο νομίζω προσφέρει μια καλύτερη επισκόπηση και καθαρή ματιά στις προτάσεις που έχει καταθέσει η Επιτροπή. Διατυπώνουμε βέβαια και κάποια ερωτήματα που θα πρέπει να συζητηθούν και να λάβουν απάντηση τους επόμενους μήνες. Είναι ενδεικτικός ο κατάλογος και όχι εξαντλητικός. Πρόκειται για μια διαδικασία νοθεώρησης που συνιστά ουσιαστικό κομμάτι αυτής της ε, βουλευτικής περίοδου. Θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, ταχαίως αλλά όχι βεβαιασμένα, να κοιτάξουμε ποιες είναι οι επικαλύψεις σε σχέση με άλλες νομοθετικές διαδικασίες όπως με δύο και ΠΕΠ. Θέλουμε να έχουμε μια γενική απεικόνηση των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και με βάση τις τομεακές νομοθεσίες και με βάση την εντολή και τις προτάσεις που έχουν ξεκινήσει από δική μας πρωτοβουλία. Επτά χρόνια μετά την εγκαθίδρυση των εποπτικών αρχών μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συλλέξει αρκετή εμπειρία Επιδιώκουμε σαφήνεια, διευκρινήσεις και επιλογές συγκεκριμένε που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το 2010, που ήμουν ήδη μέλος της Επιτροπής μας, είχα λάβει μέρος και στη διαπραγματευτική ομάδα που οδήγησε στην εγκαθίδρυση των εποπτικών αρχών. Έκτοτε βέβαια έχουν, έχει κυλήσει πολύ νερό είναι πολύ πιο περίπλοκη, πολύ η νομοθεσία. Πολλές αρμοδιότητες έχουν περάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις τράπεζες, στην εποπτεία των αγορών περισσότερο, λιγότερο στις ασφαλίσεις. Ωστόσο, σαφές είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για μια επιδίωξη κεντρικής οργάνωσης των ε, αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα στη συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Αυτή η συνεργασία και η συνεργασία και σε διεθνές επίπεδο θα συμπληρώσω γίνεται πιο περίπλοκη. Πολλές φορές ταυτόχρονα είναι πιο δύσκολο να ε, αξιολογηθεί και να ελεγχθεί. Έχουμε κάνει πολλές φορές ε, προτάσεις. Το 2015, παραδείγματι, είχαμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και τις προκλήσεις που αυτή φέρνει. Και τώρα, για να συζητήσουμε τα θέματα των ε, αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών, θα ήθελα να δώσω κάποια, κάποιες προτάσεις συγκεκριμένε, κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, βελτίωση στην ε, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δυνατότητα αξιολόγησης ε, της νομοθεσίας, ώστε αυτή να φέρνει μόνιμα αποτελέσματα, ε, κατεξουδότηση συμπράξης, τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και στον έλεγχο πάλι χρειάζεται να επισημάνουμε ότι έχει δοθεί η ερμηνεία και η διεύρυνση των εντολών δράσεως αυτών των επιτροπών, των αρχών, και επίσης ε, είναι πολύ σημαντική και έχει αποδεχθεί σημαντική η τήρηση προθεσμιών σε σχέση με τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα και την ε, ταχεία διεκπαιρέωσή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις νομοθετικές της προτάσεις δεν πραγματοποίησε ε, καμία ρηξικέλευθη κίνηση, δεν πρόκειται για επανάσταση, ούτε εμείς στο Κοινοβούλιο θα κάνουμε την επιλογή της επανάστασης για τις ε, εποπτικές αρχές οπωσδήποτε δεν πρόκειται αυτές να ανατραπούν ε, ή να αναδιατυπωθούν ε, ριζικά ούτε άλλωστε και οι αρμοδιότητές τους. Υπήρχαν και για εύστοχους λόγους τρεις διαφορετικές εποπτικές αρχές έτσι ιδρύθηκαν για λόγους σοβαρούς όπως είπα που εξακολουθούν να ισχύουν και οι τρεις τομείς ασφαλίσεις και συντάξεις, τράπεζες, αγορές είναι διαφορετικοί, διαφορετικοί τομείς με διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας και τομείς επίσης που προϋποθέτουν διαφορετικές γνώσεις και εξειδίκευση. Πρόκειται για τρεις τομείς όπου οι εποπτικές αρχές έχουν ακολουθήσει διαφορετική εξέλιξη με την άμεση εποπτική δραστηριότητα. Οι υφιστάμενες δομές πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές, να βελτιωθούν και έτσι η νομοθέτηση, η ρυθμιστική διαδικασία με την, από την εποπτική θα πρέπει να παραμείνουν διακριτές. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι σαφές ότι και η ισορροπία εξουσιών η διάκριση των αρμοδιοτήτων όπως τα λέγαμε πρέπει να είναι σαφής και η θέσπιση ενός εκτελεκτιστικού συμβουλίου το οποίο θα μπορεί να κατανέμει αρμοδιότητες δεν είναι αυτό που τουλάχιστον εγώ θεωρώ σωστή ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων. Για μένα και τις προτεραιότητες που βλέπω θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτα απ' όλα πώς μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα πιο αποτελεσματικά η νομοθεσία. Ήμουν μάλιστα επικεφαλής σε ένα τριμερή διάλογο όπου μας απασχόληθε ε, το ζήτημα των ε, πινάκων ε, υλοποίησης των λεγόμενων δισταυρούμενων πινάκων. Είχα αγωνιστεί γι' αυτό. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία που μας δείχνουν ότι δεν εξετάζεται επαρκώς η όποια παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτητα σε κάποιες λύσεις και στο σημείο αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι δραστηριότητες των υποπτικών αρχών. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι αυτή της αναλογικότητας για μένα. Η αναλογικότητα δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μεμονωμένα μέτρα, αλλά πρέπει να αποτελεί και αυτό σε αυτό συμφωνούμε όλοι πιστεύω σε μια συνολική προσέγγιση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Το βλέπουμε και στον ε, διάλογο που είναι εν εξελίξη τώρα στις προτάσεις για τις ε, τράπεζες CRR και CRD όπου ιδιαίτερα έχει αναλάβει δράση για την ομολογικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια προσέγγιση λοιπόν την οποία πρέπει να ε, στην οποία πρέπει να δώσουμε ζωή. Αυτό είναι σαφής εντολή μας και καθήκον δικό μας. Και στον τομέα των εποπτικών αρχών έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας, αλλά ε, και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Θυμούμε πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει στις διαπραγματεύσεις του 2010 να γίνουν ε, ε, διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρμοδιότητες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι ε, μια διεκδίκηση την οποία πρέπει να επιδιώξουμε ακόμη. Υπάρχουν αποφάσεις που έχουν ληφθεί χωρίς διαφάνεια και ασφαλώς αυτό είναι ένα σημείο επίκρισης το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω ότι χωρίς να έχω εξαντλήσει το θέμα και να έχω καταλήξει κάπου, έχω κάποιες ακόμη προτάσεις. Ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και ανεξαρτήτως των γεωγραφικών προτιμήσεων για, την επαν... για τον επαναπροσδορισμό της έδρας της αρχής τραπεζών που είναι λογικό να έχει κανείς γεωγραφικές προτιμήσεις, θέλω να επικρίνω την διαδικασία μέσα στην ε, συναπόφαση που πρέπει να είναι η νομοθετική διαδικασία και που δεν έχει γίνει σεβαστή από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, δεν έχει γίνει σεβαστός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Αυτό είναι λυπηρό. Και νομίζω ότι δεν αντιστοιχεί στις συνθήκες που προξενούν οι διάφορες εξελίξεις περιλαμβανομένου του Brexit. Πρέπει οι σοβαρές αυτές αποφάσεις, οι σημαντικές αυτές αποφάσεις να λαμβάνονται με σεβασμό της ε, νομοθετικής διαδικασίας. Γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε, να εξηγήσουμε στον πολίτη πώς λαμβάνουμε τις αποφάσεις, ότι λαμβάνουμε την ε, συνήθινη νομοθετική διαδικασία. Και οι πτυχές είναι οι εξής. θα ε, μεταφερθεί στο Παρίσι από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ενωθεί με την ΕΣΜΑ. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους και δίνω το λόγο στην συνεισηγήτρια και προσωρινή πρόεδρο η οποία ασφαλώς θα δώσει το λόγο στον εαυτό της. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνεισηγητά που με βοηθήσατε σε αυτή τη μετάβαση και μου δώσατε το λόγο για να σχολιάσω και εγώ. Τα έγγραφα εργασίας έχουν μοιραστεί ήδη από χθε τους συναδέλφους, οπότε φαντάζομαι πως έχουν εξοικειωθεί μαζί τους. Είναι ένα σχέδιο εργασίας αρκετά περιγραφικό. Δεν νομίζω ότι περιγράφει κάποια συγκεκριμένη θέση απριόρια, αλλά απλώς περιγράφει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θίγει και μία σειρά από ερωτήματα τα οποία προφανώς βρίσκονται και στην καρδιά της δικής μας συζήτησης. Είμαστε με τον Μπούρκαρτ Μπάλτς στην αρχή, οπότε έχουμε πολύ μεγάλο πλούτο διαφορετικών απόψεων που ακούγονται και προσπαθώ και εγώ να κάνω τη μικρή μου συνεισφορά να δώσω και εγώ το δικό μου χρώμα στην εξέταση αυτού του τόσο σημαντικού φακέλου. Γιατί όσο οδηγία και νομοθετικό κείμενο είναι ένα κείμενο σημαντικό. Θέλω καταρχήν να περιγράψω και πάλι σε ποιες συνθήκες βρισκόμαστε. Οι εποπτικές αρχές της Ευρώπης διορίστηκαν κατά τη διάρκεια μια τελείω διαφορετική συγκυρία από αυτήν στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Έχουν περάσει 7 χρόνια και στο διάστημα αυτό θα μπορούσα να αναφερθώ αυθαίρετα ίσως αλλά όχι τελείως σε τουλάχιστον τρία γεγονότα τα οποία ταρακούνησαν το τοπίο ή θα μπορούσαν να το έχουν κάνει. Καταρχήν, Τραπεζική Ένωση που οδήγησε στην δημιουργία του μηχανισμού και που στις ε, αγορές χρηματοπιστωτικές έβαλε ένα τελείως καινούριο στοιχείο από το οποίο εμείς πρέπει να διδαχθούμε κάτι. Να δούμε τι πρόοδος σημειώθηκε και πώς θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε και να δούμε τι συμβαίνει και με τις αρχές οι οποίες ε, αρχικά όχι ακριβώς δημιουργήθηκαν γιατί θα μπορούσα να πω ότι ήταν και κληρονόμοι κάποιων προϋπαρχουσών επιτροπών αλλά το δεύτερο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι η αγορά κεφαλαίων. Η Ένωση λοιπόν Κεφαλαίου Αγορών τι συνέβη όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια λευκή βίβλο αυτό το οποίο έπρεπε να είναι η έννοια κεφαλαίου αγορών, ένα γεγονός πολύ σημαντικό και το οποίο είχαμε υπογραμμίσει εμάς τότε στο ψήφισμά μας, δυστυχώς δεν είχε συνοδευτεί με μεγαλύτερη ένταξη ολοκλήρωση των εποπτικών μηχανισμών. Κάτι το οποίο είχαμε τονίσει εμείς πως πρέπει να συμβεί. Έκτοτε έχει εξελιχθεί κάπως η κατάσταση και κατανοώ ε, το γεγονός πως έχουν ξαναξεκινήσει οι προβληματισμοί. Και το τρίτο γεγονός το οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι το Brexit, λυπηρό. Το οποίο είναι ένα στοιχείο αποφασιστικό για όλους αυτούς τους φακέλους. Όταν κοιτά κανείς το έγγραφο διαβούλευσης το οποίο έβαλε στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν παρουσιάσει τις ε, προτάσεις αυτές αναθεώρησης των ιδρυτικών κειμένων νομίζω είχε ως σκοπό να προχωρήσει σε μια αναθεώρηση της όλης αρχιτεκτονικής με τις υπηρεσίες και τα λοιπά, κάτι το οποίο είχαμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο για να δούμε για όλες αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες ποια είναι η σωστή δομή. Μία αναμερίδιο αγορά, μία ολόκληρη ή να ακολουθήσουμε και το μοντέλο των δίδυμων πύργων, τα twin peaks που έχουμε σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν έκανε την επιλογή αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτό και δεν μπορώ βέβαια εγώ να εκφραστώ εκ μέρους της Κομισιόν, αλλά μου φαίνεται πως ο λόγος για τον οποίο τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε αυτή την επιλογή είναι, και αυτό έχει να κάνει και με τις αποκρίσεις ε, των όσων απάντησαν στη διαβούλευση, αλλά ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι είχαν αποφασίσει πως είχε φτάσει η στιγμή να ξεκινήσει μια απαραίτητη αναθεώρηση όχι μόνο της λειτουργίας αυτών των υπηρεσιών αλλά και κάποιων ακόμα στοιχείων οπότε και δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά λέμαργοι και ελπίζω με τον τρόπο αυτό να μην ενοχλώ κανέναν, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο τι μπορούμε να πετύχουμε στη διάρκεια αυτής της θητείας. Τουλάχιστον έτσι έχω αναγνώσει εγώ αυτή την πρόταση και πρέπει να σα πω ότι αυτό με ικανοποίησε. Κάποιοι από εσά θα θυμούνται πω πριν να βάλει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτάσει αυτέ, είχαμε την ευκαιρία να οργανώσουμε μια ανταλλαγή απόψε με τον Ζακ Ντελαροζιέρ, ο οποίο είχε επιμείνει πολύ στην τοποθέτησή του για την ανάγκη που υπάρχει να προχωρήσουμε στον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίε και να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της λειτουργίας του ω ρυθμιστικέ αρχές και της λειτουργίας τους ως εποπτικέ αρχές. Και νομίζω ότι αυτό είναι, ε, είναι μια ε, γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε ως συνεκτικό ιστό και στην ανάγνωση των κειμένων. Τώρα για τις τρεις αρχές τις εποπτικές να σας πω πως καθένα από τα κείμενα ακολουθεί λίγος πολύ την ίδια δομή, χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Είναι η... το πεδίο επέμβαση, παρέμβασης, η διακυβέρνηση και η χρηματοδότηση. Για το πεδίο. Λαμβάνουμε υπόψη τι νομοθεσία και έχει τεθεί σε εφαρμογή από τότε που δημιουργήθηκαν αυτές οι υπηρεσίες, οι πρώην επιτροπές, αλλά υπάρχουν και δύο κείμενα στα οποία αναφέρθηκε ο Μπουρκαρτ Μπάλς, κατοπινά και τα οποία δεν έχουν ε, ακόμα ε, ενταχθεί στο πεδίο το οποίο καλύπτει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα οποία νομίζω εμείς είμαστε οι αρμόδιοι. Είναι η σύνδεση με την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Σύνταξη, το περίφημο αυτό θέμα και το ΦΕΜΙΡ 2, τον κανονισμό δηλαδή για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που μιλά για τη διακυβέρνηση και την εποπτεία, όπως επίσης για τις αποζημιώσεις. Και νομίζω ότι μεταξύ αυτών των δύο φακέλων θα πρέπει να οργανώσουμε κάποιο είδους ε, αλληλενημέρωσης. Τώρα, για να τα πω και πιο επιγραμματικά, έχουμε συζητήσει με τις αρμόδιες αρχές Και πρέπει να σας πω πως, αν κατάλαβα καλά, έχουμε πολλές καταγγελίες και παράπονα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή στη διαδικασία λήψης απόφασης με τρόπο που αυτές οι αποφάσεις να είναι αποτελεσματικές. Ξεκινώντας από αυτή τη διαπίστωση, θα έλεγα πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μία πρόταση η οποία εμπνέεται από άλλα ε, είδη διακυβέρνησης με ένα executive board, ένα εκτελεστικό συμβούλιο, στο οποίο θα επανέλθουμε. Θα κάνουμε προτάσεις και τροποποιήσεις, αλλά ξεκινάμε εδώ από την αρχή την πεποίθηση πώς. Και πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά. Οι εθνικές αρχές, οι εποπτικές, οι ελεγκτικές, οι οποίες ουσιαστικά εκπροσωπούνται σε αυτό το εποπτικό συμβούλιο, εκπροσωπούν τα εθνικά του συμφέροντα. Αυτά γνωρίζουν και έχουν μια προσθεμένη αξία και συνεισφέρουν με τον τρόπο αυτό ε, από κοντά, με πραγματογνωμοσύνη. Όμως, όταν χρειάζεται να τροποποιήσουμε νομοθεσία, το κίνητρο να αλλάξουν τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος διατήρησης του status quo ή συντηρητισμού και αυτό φαίνεται και στον απολογισμό που κάναμε και είπαμε πως αυτό θα πρέπει να το ξεκινήσουμε περάσουμε. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και η ιδέα αυτού του Executive Board. Τώρα για τον τρόπο χρηματοδότησης, δεδομένων των περιορισμών που έχει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, δεν μπορεί να συνεισφέρει πάνω από το 40% της χρηματοδότησης αυτών των υπηρεσιών και εκεί βεβαίως υπάρχει ανησυχία γιατί με τον τρόπο αυτό, όπως μας είπαν και οι παίκτες στην αγορά, μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα, μια αυξητική τάση στους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών, οπότε θα πρέπει να διατηρηθούν αυτοί μέσα σε λογικά πλαίσια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στα οποία θα μπορέσουμε να επανέλθουμε και να πω μόνο δύο λόγια για την Επιτροπή για τους Συστημικούς Κινδύνους, γιατί πιστεύουμε εφόσον στην πρόταση δεν ξανανοίγουμε την αρχιτεκτονική όλων των υπηρεσιών, πιστεύω πως το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και για την περίπτωση αυτής της Επιτροπής. Για να είμαι πλήρης πρέπει να σας πω πως έχει τη βούληση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβουμε στη διακυβέρνηση των υπηρεσιών στόχους πιο ταυτοποιήσιμους Εποπτεία, ρύθμιση, καινοτομία για τα καινούργια χρηματοπιστωτικά, τα fintech όπως τα ονομάζουμε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την προστασία του καταναλωτή. Και θα κλείσω λέγοντας απλώς πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη γνώμη του πιστεύει πως θα πρέπει να ενισχύσουμε την πρόταση αυτή γιατί εμείς βεβαίως θα ε, διορίσουμε και εμείς, ε, θα είμαστε μέλος της διαδικασίας για το διορισμό των μελών αυτού του Executive Board, αλλά θα πρέπει να μην αφήσουμε στην άκρη θέματα όπως η προστασία του καταναλωτή, γιατί και εκεί πιστεύω πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τα όσα υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι. Έκλεισα λοιπόν τη δική μου παρέμβαση και με έκοψε η πρόεδρος. Και γι' αυτό ως πρόεδρος τώρα δίνω το λόγο στην ECR για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συνηγητές ε, για το πολύ χρήσιμο εγγραφό εργασία το οποίο διανεμήθηκε σε εμά και το οποίο είχα τη δυνατότητα να ε, διαβάσω μία μόνο φορά, αλλά θα χρειαστεί να το διαβάσω περισσότερες φορές ούτως ώστε να, μπορώ να, να μπορέσω να αντιληφθώ όλα τα ερωτήματα που θέλετε εκεί. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω στα ερωτήματα που θέσατε στο τέλος αυτού του εγγράφου. Αλλά επιτρέψτε μου αρχικά να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Το έγγραφο επανεξετάζει και την αρχή της όλης διαδικασίας ε, και αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο αρχικά δημιουργήσαμε τις ευρωπαϊκές ε, εποπτικές αρχές, ε, οι οποίες δεν ήταν ίδιες μεταξύ τους, ε, παρότι παρόμοιες ε, και πράγματι τώρα στο ενδιάμεσο διάστημα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά οι τρεις ε, διαφορετικές αρχές και σε ό,τι αφορά τις, τις αρμοδιότητές τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τον τομέα στον οποίο εστιάζουν και νομίζω πως αυτό είναι, ήταν αναμενόμενο, οπότε θα πρέπει να τις εξετάσουμε και διαφορετικά όταν θα περάσουμε στην πανεξέταση τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που θέσατε προς συζήτηση σε ό,τι αφορά τι ε, αξιολογήσει αντικτύπου, πράγματι έχετε δίκιο. Πάντοτε εμεί δηλαδή ανέκαθεν λέμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου ότι χρειαζόμαστε ρεαλιστική προσέγγιση και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε αξιολογήσει αντικτύπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ερώτηση ε, 50 ε, και την σχέση με τις ECA, ναι, νομίζω πω θα πρέπει να εστιάσουμε ειδικότερα σε αυτό το τομέα. Ε, Εμεί ε, από τη ε, δική μου πλευρά πάντοτε είμαστε υπέρ ενό ισχυρού ρόλου των εθνικών αρμοδίων αρχών προκειμένου να σεβαστούμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Οι αγορές δηλαδή των κρατών μελών που ορισμένες φορές βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους λόγω ακριβώς της εμπειρογνωμοσύνης που έχουν συγκεντρώσει οι αποπτικές αρχές, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη των διαφορετικών κρατών μελών. Επίση, ό,τι αφορά το σημείο 38 ε, και το ερώτημα που μα έχετε θέσει ω προ το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε την, ε, και την, να βελτιώσουμε την εφαρμογή τη ενωσιακή ε, νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Νομίζω πω αυτό το κατέδειξε η MIFID 2, όπου δεν είδαμε δηλαδή εφαρμογή περίπου στο ίμιση των κρατομελών και αυτό από την 3η Ιανουαρίου. Έω την 3η Ιανουαρίου του 2018 λοιπόν τα, τα μισα κάτι κράτη-μέλη δεν το έχουν εφαρμόσει και εκείνα που το έχουν κάνει δεν το έχουν κάνει με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, και από εκεί και μετά τίθεται το ζήτημα ε, της, της σχέσης μεταξύ αυτών των, ε, ε, ε αυτών των αρμοδιοτήτων και των εποπτικών αρμοδιοτήτων. Και εγώ δεν είμαι πεπισμένη. Δηλαδή χρειαζόμαστε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την κατάλληλη νόμο παραγωγή και βέβαια προϋποθέτει κάτι τέτοιο και μια εις βάθος γνώση ε, της αγοράς και των φορέων της αγοράς. αυτή λοιπόν η, γνώση ε, συγκεντρώνεται μέσω της εποπτείας της αγοράς, οπότε δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα συνέχεια, συνέχειας, συνέπειας αν θέλετε, ένα ζήτημα που, στο οποίο θα επανέλθω, ε, εδώ αναφέρομαι ειδικότερα ε, στο σημείο 48 και τη σχέση μεταξύ ΕΜΙΡ και ΠΕΠ. συμφωνώ με αυτό που λένε οι συγητές, ότι δηλαδή θα πρέπει να εξετάσουμε και την σχέση την ε, συνέπεια μεταξύ των διαφορετικών ε, προϊόντων ε, και πώ μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ IDD και MIFID 2. Εδώ έχουμε δηλαδή πολύ παρόμοια προϊόντα, τα οποία όμως ε, ουσιαστικά υπάγονται σε διαφορετικά, διαφορετικές δέσμες κανόνων, ενώ προορίζονται για τους ίδιους καταναλωτές. Μήπως χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ περισσότερη συνέπεια σε ό,τι αφορά τα όσα προβλέπουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την περισσότερη συγκέντρωση ε, των αρμοδιοτήτων στην σας, ναι, θα μπορούσαν να παίξουν ενισχυμένο ρόλο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την οδηγία MIFID, πάντοτε λέγαμε στην δική μας Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενοποιημένη προσέγγιση ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, την ε, διάθεση των σχετικών πληροφοριών, σε ό,τι αφορά τις ε, σχετικές συναλλαγές. Σε 15 λεπτά αφότου έχει δοθεί η εντολή της ειδικότερα στους τομείς ΕΦΙΝΤΑ και VECTEC, κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε, ούτως ώστε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και θα βοηθούσε και τους επενδυτές σε ό,τι αφορά τη λήψη των αποφάσεών τους. Όμως ε, δεν ξέρω ε, κατά πόσο θα προκύψει μια εμπορικού χαρακτήρα λύση για κάτι τέτοιο, αλλά ίσως η ΕΣΜΑ εδώ θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε δηλαδή να κάνει κάτι προς όφελος των καταναλωτών της ε, Ένωσης. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να αναλάβει μια ευρύτερη αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα και των πληροφοριών η ΕΣΜΑ. Υπάρχουν από εκεί και μετά μια σειρά αποζητήματα σε ό,τι αφορά τι τις ε, εποπτικές αρχές, τα διεθνή όργανα τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ε, διάφορες ε, συμφωνίες και αποφάσεις ισοδυναμίας. Πάντως, εκείνο που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι οι αποφάσεις ισοδυναμίας αυτή τη στιγμή με τον τρόπο δηλαδή που λαμβάνονται είναι πολιτικού χαρακτήρα και λαμβάνονται από την Επιτροπή. Και μια σειρά από τέτοιες αποφάσεις ήταν ουσιαστικά πολύ αρνητικέ σε ό,τι αφορά την, το κύρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ό,τι αφορά την που να προβλέπει το πώ θα αντιμετωπίζουμε του άλλου παίκτε παγκοσμίω ε, και αν του διαφοροποιούμε, με βάση ποια κριτήρια του διαφοροποιούμε. Άρα λοιπόν αυτό που μας προτείνει τώρα η ε, Επιτροπή είναι να βασίζουμε αυτή την αναγνώριση της ισοδυναμίας στην σημασία των υπολείπων ε, περιοχών του πλανήτη και όχι να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αν συνδυάσουμε λοιπόν αυτή την προσέγγιση με την προθεσμία των 30 ε, ημερών, ουσιαστικά το αποτέλεσμά του είναι αρνητικός αντίκτυπος στη για επενδύσεις εντός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως ακριβώς οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές μπορούν να μας βοηθήσουν εδώ να βελτιώσουμε το κλίμα. Δηλαδή με τέτοιου είδου εργαλεία εποπτείας παρακολούθησης ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μια αντιστάθμιση σε ό,τι αφορά τον αρχηγό αυτών των αποφάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κλίντ, εκ μέρου των Φιλελευθέρων. Πρόεδρε, οι πέντε πρόεδροι στην έκθεσή του για την ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση τον Ιούνιο του 2015 ζήτησαν να υπάρχει ε, μια ενιαία ε, εποπτική αρχή για την ενιαία αγορά. Μπορεί αυτό να σας φαίνεται απλό, αλλά μεταφραζόμενο στα γερμανικά καταλήγει σε αποτέλεσμα άλλο από αυτό που θα καταλάβαινε κάποια άλλη, κάποια άλλη γλώσσα. Δηλαδή στα γερμανικά θα σήμαινε ενιαία αρχή εποπτείας της αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την αγορά, την κεφαλαία αγορά. Τότε θα πρέπει να υπάρχει εποπτική αρχή που θα αποτρέπει τις συνεννοήσεις και που θα οδηγεί σε μια ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας. Αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής. Μπαίνει προς την ορθή κατεύθυνση. Με βάση αυτή πρέπει να συζητήσουμε και να την βελτιώσουμε βεβαίω. Μέχρι τώρα οι τρεις εποπτικές αρχές έχουν κάνει αξιόλογη δουλειά δεν μπορεί να ισχυριστεί κανεί δηλαδή ότι πρέπει να ανατραπεί το σύστημα γιατί έχουν αποτύχει. Για, για το τεστ αντοχή των τραπεζών, βέβαια μπορεί να μην ήταν επιτυχέ το πρώτο τεστ αντοχή που έκανε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Η Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Συνταξιδοτικών Ταμείων δεν έχει καόσα θα μπορούσε να έχει κάνει. ΔΕΣΜΑ έχει κάνει καλή δουλειά και για τους ε, οργανισμούς αξιολόγησης επιστολυπτικής ικανότητας και για τα ρέπος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να κοιτάξουμε την ε, διαχείριση, την ε, χρηματοδότηση, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εδώ νομίζω οι αρμοδιοτήτες θα είναι το σημείο στο οποίο θα κρυθούν τα πάντα. Οι διαχωριστικές γραμμές βεβαίω μεταξύ των εθνικών και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οπωσδήποτε δεν πρέπει οι εθνικές εποπτικές αρχές να θεωρήσουν ότι αντιμετωπίζονται ως αρχές δεύτερης κατηγορίας και άρα να ε, χάσουν το ενδιαφέρον τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να συμβάλλουν χάρη στις γνώσεις τους πάρα πολύ στο εποπτικό αυτό έργο και πρέπει να βρουν τη θέση τους ε, ε, μέσα στο νέο αυτό σύστημα για να μην υπομονωμευθεί. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα, να υπάρχει σαφής ε, διαφοροποίηση, διάκριση των εξουσιών και ε, μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και από αυτό θα κριθεί και η επιτυχία του νέου συστήματος. Βεβαίως με κάποιο τρόπο θα πρέπει να καθοδηγούν τις εθνικές αρχές οι ευρωπαϊκές χωρίς όμως από εξέδρας ε, επιβολή όρων και ε, παρακολούθησης. Εάν έχουμε ένα εκτελεστικό συμβούλιο, το βρίσκω, βρίσκω καλό, πρέπει όμως να είναι αποτελεσματικός ο εποπτικός φορέας. Πόσα μέλη θα έχει, 5, 3, 2, περισσότερα, λιγότερα, δεν είναι οπωσδήποτε το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο είναι να κάνει τη δουλειά του αυτό το Συμβούλιο ε, αποτελεσματικά, όπως επισημαίνεται και εδώ, με ε, τακτικέ συναντήσει. Γιατί εδώ αναφέρεται ότι έχει πέντε φορές το χρόνο συνάντηση. Με αυτό δεν μπορεί να κάνει ουσιαστική εποπτική δουλειά. Μια φορά το μήνα τουλάχιστον, αν όχι περισσότερο, και με προετοιμασία του ε, Γενικού Συμβουλίου των Εποπτικών Αρχών. Έτσι μπορεί να κάνει πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική δουλειά. Για το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου λυπούμαστε που δεν έχει καλύτερη εκπροσώπηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εποπτικές αρχές δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου, ούτε υπεράνω του πολίτη και άρα είναι υποχρεωμένες σε λογοδοσία. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ρόλο του ως όργανο στην υπόθεση αυτή. Χρηματοδότηση. Ξέρω ότι έχει περιορισμού ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, πάνω από 40% δεν μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το να λέμε ότι τα υπόλοιπα πόσα καλύπτονται από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι υπερβολικό πιστεύω. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κατανομή 40-30-40 20-20-20 βεβαιως και οι εθνικές αρχές θα παίρνουν χρήματα από, τον, από τον κλάδο το χρηματοπιστωτικό αλλά σημασία έχει εδώ να διατηρηθούν μέσα στο παιχνίδι να μην αποκλειστούν οι εθνικές αρχές και να μην θεωρήσουμε ότι ανοίγουμε την κάνουλα και τρέχει χρήμα. Πρέπει να είναι αποτελεσματική η χρήση των κονδυλίων. Η ενσωμάτωση δε περιβαλλοντικών, κοινωνικών και άλλων πτυχών δεν με βρίσκει αντίθετο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επαλήθευση και την υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων. Ωστόσο, βιώσιμη επένδυση σημαίνει ταυτόχρονα και σταθερή Μπορεί να είναι πράσινη μια επένδυση, αλλά να, ε, έχει, να φέρει υψηλό κίνδυνο. Να μην στηρίζεται σε τεχνολογικές εξελίξεις και άρα να μην είναι σταθερή. Σε αυτό θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εν κατακλείδη πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Πρόεδρος, θέλετε να καταλήξετε. Ναι, ναι, Πρόεδρε, καταλήγω στα συμπεράσματα. Ε, πιστεύω ότι θα χρειαστεί ε, πολύ λεπτομερή συζήτηση και με τις εθνικές αρχές και με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και με το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόεδρο Συγκούε, δεν εκπροσωπείται. Θα παρακαλέσω τον Σβέν Κίγκολτ να λάβει το λόγο και ζητώ συγγνώμη διότι θα έπρεπε στην αρχική μου παρέμβαση να επισημάνω ότι οι εργασίες του Κοινοβουλίου που αποτελούν και τη βάση εξέτασης ε, αυτής της νομοθεσίας στηρίζονται και βέβαια στο ψήφισμα για την ενώση των κεφαλαίων αλλά και στις εργασίες της προηγούμενης ε, βουλευτικής περίοδου όταν εσείς κύριε Γκίγκολτ ήσασταν εισηγητής και είχατε μιλήσει για το σχεδιασμό αυτών των ε, υπηρεσιών, των αρχών. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό το σχόλιο. Έχουμε προϊστορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε αυτές τις εποπτικές αρχές να γίνουν πιο ευρωπαϊκές, πιο αποτελεσματικές και να δρουν και με ένα λογικό τρόπο. Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν η βασική ιδέα και θυμάμαι πολλές νύχτες με τριμερή διάλογο για να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Έχουμε κάνει πολύ θετικές αλλαγές. Γιατί, Γιατί έχουμε αυτό το κοινό όραμα. Και ελπίζω πως το όραμα αυτό θα μας οδηγήσει σε μια ενιαία αγορά κεφαλαίου αγορών όπου οι καταναλωτές και οι επενδυτές θα συμβιώνουν στα πλαίσια του κοινού μας οράματος και θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι καταφέραμε, τι πετύχαμε, πού κάναμε λάθος και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη από αυτή από την οποία προερχόμαστε που ήταν ο ρυθμιστικός ανταγωνισμός χωρίς να υπάρχει μεγάλος βαθμός ολοκλήρωσης αγοράς και η Ευρωζώνη μας αποδεικνύει σαφέστατα γιατί του υπάρχει μακροοικονομική ανάγκη για περισσότερο ε, ολοκληρωμένες ε, κεφαλαίου Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πορεία και από τη δική μου έκθεση του 2014, μετά από πάρα πολλή συζήτηση μεταξύ μας, βοήθησε στο να επηρεάσουμε τουλάχιστον εν μέρη, πρέπει να είμαστε μετρημένοι στα όσα λέμε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις που κατέθεσε και ένα από τα στοιχεία κλειδιά στα οποία, τα οποία διαπιστώσαμε είναι πως αυτές οι αρχές δεν έχουν χρησιμοποιήσει όλες τις αρμοδιότητες με τις οποίες έχουν πρικοδοτηθεί. Γιατί. Γιατί οι αρχές των κρατών μελών που είναι απαραίτητες για κάθε σχετική απόφαση δεν θέλουν να ελέγξουν η μία την άλλη γιατί ξέρουν ότι αν ελέγξουν κάποιον άλλον τότε μπορεί να είναι οι επόμενες που θα ελεγχθούν και βέβαια αυτά όλα δυσκολεύουν την ε, κατάσταση. Οπότε ο φυσικός ρόλος του Κοινοβουλίου εδώ είναι να υπερασπιστεί και να διευρύνει αυτά τα μετρημένα βήματα τα οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτές τις ε, αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πιο ευρωπαϊκές και να δομηθούν με έναν τρόπο που θα υπάρχει περιορισμός στη σύγκρουση συμφερόντων και κάτι το οποίο δεν καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό όταν τις δημιουργήσαμε είναι να εξετάσουμε σε βάθος στο τι θα γίνει με το μακροπροληπτικό ε, κομμάτι της εποπτείας. Του είπε ο Μπόρχαρτ, η ενδυνάμει σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει και στα πλαίσια της ίδιας της ΕΚΤ και πρέπει να σας πω ότι σε κάποια, στην περίπτωση της Τραπεζικής Ένωσης έχουμε ε, και άτομα των οποίων η καριέρα εξαρτάται από το αν η ε, μακροεποπτεία πέτυχε, εάν προβλέψαμε τις κρίσεις ή όχι και υπάρχει ένα τεράστιο σώμα, ένας φορέας, ο οποίος επιτρέπει σε όλους να μην είναι υπεύθυνοι στην περίπτωση που οι προβλέψεις θα πέσουν έξω. Εν πάση πρέπει να σας πω ότι αυτή η διακυβέρνηση να ανισχύει περισσότερο από αυτές ε, των εποπτικών αρχών. Γιατί όταν τις δημιουργήσαμε, τις συμπληρώσαμε με κάποια σημαντικά στοιχεία για την προστασία των επενδυτών, για την προστασία των καταναλωτών. Αυτά βρίσκονται στην εντολή τους, αλλά δεν αλλάξαμε τουλάχιστον με ουσιαστικό τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το προσωπικό τους. Οπότε προσθέσαμε αρμοδιότητες, αλλά δεν προσθέσαμε προσωπικό. Και βέβαια, εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε τους προϋπολογισμούς. Τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στο θέμα αυτό και χαιρετίζω τα όσα είπε η συνάδελφος και η Σουίνμπορν και αυτά τα έχετε βάλει και στην έκθεσή για την απαλλαγή για να δούμε πόσος χρόνος και χρήμα χρειάζεται για ρυθμιστικές ε, διαδικασίες και πόσες για την επιβολή και για την προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών. Ο ρόλος ε, στην κοινωνική και του εργολογική επένδυση των ρυθμιστικών αρχών, ε, των εποπτικών αρχών, με συγχωρείτε, δεν είναι να λέμε ότι όποια επένδυση είναι πράσινη δεν έχει κίνδυνο. Όχι. Ο στόχος είναι αυτοί οι επενδυτές να γνωρίζουν ποια προϊόντα είναι κοινωνικά, ποια είναι περιβαλλοντολογικά και να ενημερώνονται και για τους κινδύνους που περιέχουν έτσι ώστε να λαμβάνουν μία απόφαση βασιζόμενη σε επιχειρήματα. Οπότε αν θέλει κανείς νέες τεχνολογίες, γιατί η πράσινη τεχνολογία ε, είναι πολύ πιο ε, επικίνδυνη από το να κάνει κανείς τα γνωστά και βαρετά. Γι' αυτό λοιπόν διαφάνεια, εξήγηση του πού βρίσκεται ο κίνδυνος, όχι έτσι ώστε να προωθήσουμε ε, κάποια προϊόντα ως ασφαλή, ενώ δεν είναι, και να τα προωθήσουμε, οπότε οι αρχές έχουν κάποιο ρόλο και αυτός δεν θα πρέπει να συγχαίεται με ένα ρόλο marketing, γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Καλές οι προτάσεις και νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να αναγνωρίζονται και στην τομεακή νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Catch the eye αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει το λόγο μπορεί να το ζητήσει. Κυρία Χούμπνερ έχει το λόγο. Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο τώρα με τη διαδικασία Catch the Eye. Κύριε Χέις, μόνο εσείς. Ωραία. Ντανούτα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που παρουσιάσατε αυτό το έγγραφο εργασία που μας μοιράστηκε χθε. Πολύ χρήσιμο για κάποιον σαν εμένα που είμαι άλλωστε και η συγγήτρια ε, για τον ε, κανονισμό το ΦΕΜΙΡ 2 ε, και τη σχετική γνωμοδότηση. Κάποια στιγμή πρέπει να ενισχύσουμε την αρχιτεκτονική των εποπτικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση για όλο το σύστημα. Κάτι το οποίο θα κάνει αξιόπιστες εποπτικές αρχές ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει και στην αποτελεσματική διακυβέρνηση μέσω αυτών, κυρίως στα τραπεζικά. Οπότε η ΕΣΜΑ αυτή τη στιγμή πάνω από του αντισυμβαλόμενους για παράδειγμα έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Ε, όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σε ένα ε, πολύ θετικό αποτέλεσμα που θα τη βοηθήσει να λειτουργεί καλύτερα. Να υπενθυμίσω πως χρειαζόμαστε και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών αντισυμβαλόμενων όπως και των αντισυμβαλόμενων από τρίτες χώρες και να δούμε τη συνέργεια που μπορούμε να έχουμε μεταξύ όλων αυτών των εποπτικών αρχών που μπορεί να είναι τρίτων χωρών ή ευρωπαϊκών γιατί πιστεύω πως αυτό είναι ο στόχος της πρότασης. Μόνο τότε θα καταφέρουμε οι συνέργειες αυτές του συστήματος να δώσουν καρπούς, αν δώσουμε επιπλέον πόρους, επιπλέον βοηθήματα. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν έτσι ώστε να έχουν την εποπτεία όχι μόνο των Ευρωπαίων αντισυμβαλωμένων αλλά και των αντισυμβαλωμένων τρίτων χωρών. Και νομίζω πως και οι τρίτες χώρες έχουν να κερδίσουν από αυτές τις επιπλέον αρμοδιότητες τις εποπτικές. όπως άλλωστε και οι Ευρωπαίοι. Και θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται με αυτή την ε, ακυριότητα της εποπτείας έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιφάσεις στην εφαρμογή και κυρίως να μην δημιουργήσουμε πολύπλοκα συστήματα εκεί που δεν χρειάζονται. Ο κύριος Χέιζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, και συγχαίρω σας και το μπουκάρτε για το έγγραφο που προετοιμάσατε επί το οποίο κάνουμε τη συζήτηση τώρα. Και πράγματι, αν συγκρίνουμε ε, τι θέσει μα με το που βρισκόμαστε τώρα, πράγματι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη φάση και αυτό καταδεικνύει και την εντοχή μα ε, σε γενικέ γραμμέ τη Ένωση. Ε, και βέβαια αυτή η εντοχή οφείλεται στα συστήματα που δημιουργήσαμε μετά από την κρίση και τα οποία ακριβώς κατέδειξαν αυτή την αντοχή μας και επέτρεψαν στην οικονομία της Ένωσης να ανακάμψει. Αυτά δηλαδή οφείλονται στι βελτιώσεις που επήρθαν στο κανονιστικό πλαίσιο και οποιαδήποτε αναθεώρησή του θα πρέπει να γίνει ακριβώ των θετικών στοιχείων και των αρνητικών στοιχείων εκείνων, δηλαδή που απέδειξαν την αξία του ε, στην πράξη για εκείνο που δεν το έκαναν. Πάντω, ε, σε ό,τι αφορά τι πέντε ε, πρακτικέ, είτε αφορά τον τομέα των ασφαλίσεων είτε των τραπεζικών υπηρεσιών, σίγουρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονό ότι πράγματι οι αλλαγέ τι οποίε κάναμε λειτουργήσαν σε γενικέ γραμμέ. Ναι, χωρί αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να, προβούν, να προβούμε σε αναθεώρησή του έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο λειτουργούν αποτελεσματικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση τη Επιτροπή. Ναι, πράγματι χρειάζεται για αυτή η κανονιστική διαμεσολάβηση, αν θέλετε. Γιατί θέλουμε και εμεί να αξιοποιείται πλήρω η νέα αγορά. Ε, ε, και οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε επιτρέψουν ακριβώ την ε, ολοκλήρωσή τη. αλλά εάν κινηθούμε ε, προς ένα πλήρως εναρμονισμένο σύστημα και ε, όλες οι σχετικές αρχές ε, λειτουργούν σε επίπεδο ένωσης, τότε θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα που θα δημιουργήσουμε να ανταποκρίνεται στο στόχο μας. Προφανώς δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή, αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται σε ό,τι αφορά την κανονιστική αρμοδιότητα. Σίγουρα το σύστημα που θα πρέπει να δημιουργήσουμε θα πρέπει να είναι εντάξει των περιστάσεων. Τώρα, εάν έχουμε υπερβολικά εναρμονισμένη ή πολύ εναρμονισμένη προσέγγιση, ε, τότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρηθεί ο ανοιχτό χαρακτήρα. Δεν θέλουμε έναν προστατευτισμό από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέκαθαν είμαστε ανοιχτοί σε επενδύσει ε, από την Αλοδαπή. Και αν δούμε και το τι συμβαίνει στι ΗΠΑ σε αυτή την περίοδο, σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την εισδροή επενδύσεων, ξένων επενδύσεων προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού αλλά θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά ε, ταμεία όπως ε, το και άλλα, είχαμε την δραστηριοποίηση ορισμένων τρίτων χωρίς να έχουν λάβει δηλαδή την κατάλληλη έγκριση από την ΕΣΜΑ και οπότε θα πρέπει ε, στο μέλλον η δραστηριοποίηση αυτών των χωρών να ε, υποβάλλεται σε καλύτερη ε, εξέταση και από την ΕΣΜΑ. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε ποιε είναι οι απαιτήσει οι οποίε θα αφορούν στο outsourcing και τι ισχύει σε ό,τι αφορά τι συνθήκε τη αγορά εργασία. Προφανώ προκύπτουν από εκεί και μετά κάποια ζητήματα σε συνέχεια του, του Brexit και κάτι το οποίο μα ανησυχεί ιδιαίτερα είναι αυτό τη εγχώρηση αρμοδιοτήτων. Δηλαδή, αν πραγματικά είναι πολύ σκληρό το Brexit, δεν ξέρουμε ε, κατά πόσο αυτά τα αν χαθεί το πάσπορτ δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε ήδη ε, κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός κανονισμού του προσπέκτου και βλέπουμε πως η, πρόταση, η Επιτροπή προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτή την προσέγγιση και νομίζω πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μια καλή διαδικασία παραγωγής. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε την κατάλληλη ασφάλεια και την κατάλληλη προβλεψιμότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τότε θα πρέπει να κινηθεί διαφορετικά η Επιτροπή. Και όπως είπατε και εσείς, ε, ίδια Πρόεδρε, ε, σε ό,τι αφορά τι ε, κεβαλαγορέ ε, και από εκεί και μετά το securitization και το prospectus, έχουμε κάνει πολλά. Δεν μπορούμε λοιπόν από εκεί και μετά, στο πλαίσιο αυτή τη αναθεώρηση που θα κάνουμε, να θέσουμε ακόμα ε, περισσότερε γενικότερε ε, προποθέσει και να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερο γραφειοκρατικό άχθο. Δεν αναφέρομαι βέβαια στο εποπτικό ζήτημα και το ζήτημα τη πιστοποίηση, αλλά σε ό,τι αφορά την, την, την, το να προδικάζουμε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ε, ομότητες που θα έχουμε. Δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά το δυναμικό της νομικής και νομισματικής ένωσης. Αυτά που λέω να μου ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει το λόγο. Αν όχι, δίνω το λόγο στον Μπούρχαρτ. Για να δείτε πώς θα συμπράγμαται αυτής της πρώτης ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδης ηγητές και όλους τους συναδέλφους που έλεγαν το λόγο σήμερα σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να γίνει αυτή η ανταλλαγή, το ότι γίνεται αυτή η ανταλλαγή τόσο πρώιμα στην ε, διαδικασία. Και ιδιαίτερα σήμερα πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε πώς θα εξασφαλίσουμε, θα εξακολουθήσουμε να εξασφαλίζουμε την ε, χρυσή αυτή τομή, την ισορροπία τη λεπτή μεταξύ των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών αφενός και των εθνικών εποπτικών αρχών αφετέρου. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που ο κύριος Κλίντς να μην μετατραπούν σε αρχές δεύτερης κατηγορίας ή να μην αποκομίσουν την εντύπωση ότι είναι αρχές δεύτερης κατηγορίας οι εθνικές εποπτικές αρχές. Το υπογραμμίζω και εγώ. Και επίσης στη, στην ε, παρατήρηση του άλλου συναδέλφου σε σχέση με το Σύμβουλο Συστημικού Κινδύνου και τη, διάκριση των αρμοδιοτήτων. Συμπερασματικά λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε την, ε, ε, το διαχωρισμό στην ρυθμιστική αρμοδιότητα, αφενός και την εποπτική αφετέρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα να ε, τονίσει και να συμπεριλάβει βέβαια στις συζητήσεις του. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και περιμένω την περιουτέρω συνεργασία και με σένα περιμένως και με τους λοιπούς συνεισηγητές ε, και οδησηγητές και βέβαια με τους συναδέλφους στην Επιτροπή. Κυρία Μπερές. Ευχαριστώ πολύ. Θα έπρεπε ίσως να το έχω πράξει νωρίτερα. Πρέπει να ρωτήσω αν υπάρχει εκπρόσωπος Επιτροπής που θέλει να λάβει το λόγο. Έχουμε λίγο χρόνο στη θεσή μας, χωρίς βέβαια να είναι υποχρεωτικό ε, να τοποθετηθείτε. Μια πρώτη εξέταση μόνο κάνουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Μπουρχαρτ Πάλτς για αυτήν την πρώτη ανταλλαγή, όπως επισήμανε και ο ίδιος. Σημειώνω πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για την κυρία Σουίνμπερν που επισημαίνει τις ε, ε, διαφορές ε, εκτίμησης μεταξύ των ε, διαφόρων νομοθεσιών και βεβαίως το ρόλο που θα έχουν οι εθνικές ελεγκτικές αρχές πρέπει να γίνεται αυτό σεβασμός. Εκείνες γνωρίζουν καλύτερα πώς λειτουργούν οι αγορές, έχουν εις βάθος γνώση των αγορών. Ταυτόχρονα όμως, στηριζόμενοι σε αυτή την γνώση και εξειδίκευση, πρέπει να οδηγηθούμε σε μια συνολική ε, θεώρηση ευρωπαϊκή. Και αυτή τη στιγμή η ισορροπία μεταξύ των αρχών εθνικών και ευρωπαϊκών δεν υπάρχει. Επισημάνατε και εσείς ότι δεν πρόκειται να κρυθούν οι ισοδυναμίες μέσα από την έκθεση αυτή αλλά από, την, από τις εξουσίες που έχει προσλάβει παραδείγματι η ΕΣΜΑ ε, οδηγούμε στη διατύπωση μιας πρότασης για τη ρύθμιση των ισοδυναμιών και για το μέλλον. Για τον κύριο Κλίντς, όταν λέτε ότι θα πρέπει από καθέδρας και αφιψηλού να επιβάλλονται από τις ευρωπαϊκές αρχές τις εθνικές ε, το τι θα κάνουν ναι, από την άλλη οι εθνικές αρχές δεν έχουν ρόλο να παρεμποδίσουν κάθε πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ο κίνδυνο και αυτή είναι η ισορροπία που πρέπει να αποκαταστήσουμε. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Οι εθνικές ελεγκτικές αρχές και ζητώ συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω μια κάπως ε, απλοκή έκφραση ε, κάνουν ε, ε, λίγο το παιχνίδι της κολοκυθιάς, δηλαδή σου πετάω το μπαλάκι, αν κουνηθείς εσύ σε, σε, ε, εγώ, και τελικά ακυρώνεται κάθε προσπάθεια. Χρειάζεται περισσότερη σύγκληση. Και στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικέ αρχές ελέγχου υλοποιούν την νομοθεσία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλλουν σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πνεύμα. Ο Σβέν Γκίγκολτ, όταν είπε ότι οι ελεγκτικέ αρχές δεν εξαντλούν τι εξουσίες του και τι δυνατότητε που αυτέ προβλέπουν, αυτή η, αυτό, αυτός ο αυτοπεριορισμός που υπάρχει ε, πρέπει να ξεπεραστεί πλέον. Στην διάρθρωση σε σχέση με την ε, οδηγία ΕΜΙΡ θα απαντήσω ότι ναι, όταν βλέπει κανείς πώς έχει διατυπωθεί αυτή είναι οδηγία η οποία ε, διατυπώθηκε πριν η Επιτροπή να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για τις ελεκτικές, για τις εποπτικές αρχές. Διότι στην ΕΜΙΡ 2, στον ΕΜΙΡ 2, κανονισμό ΕΜΙΡ 2, γίνεται λόγος για ε, συμβούλιο διοικητικό το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Γίνεται λόγος για διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΜΑ που δεν υπάρχει πλέον, δεν προβλέπεται στην αναθεώρηση ε, τη ΕΣΜΑ όπως αυτή προτείνεται. Επομένω και εμείς έχουμε εκεί να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, συνεχίζοντας τη σκέψη του Μπουρκάρτ Μπάλτς, Λυπούμε που εμείς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, αντιλαμβανόμενοι ότι το Συμβούλιο είχε αρχίσει να αναπτύσσει μια συζήτηση για τα κριτήρια με βάση τα οποία θα κρίναμε την ε, αλλαγή της έδρας των υπηρεσιών δεν δραστηριοποιηθήκαμε επαρκώς. Συμβαίνει πολλές φορές να κάνουμε προκαταρκτική συζήτηση σε θέματα που έχουμε αρμοδιότητα ως νομοθέτες και αυτό θα έπρεπε να είχαμε κάνει αντί να περιμένουμε να γίνει αυτή η επική μάχη ε, για τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής, Τράπεζας, Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Εποπτείας των Τραπεζών και το κόστος του ενοικίου για τα νέα της κτίρια αντί να έχουμε δώσει εμείς συγκεκριμένε προτάσεις και άλλα κριτήρια για την επανεγκατάσταση της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Καλό θα είναι λοιπόν να επισημάνουμε στο Συμβούλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη τελικά η απόφαση δεν ε, σέβεται τα, ε, τις εξουσίες του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Χρονοδιάγραμμα τώρα για την εξέταση της πρότασης. Ξέρω ότι ήδη έχετε πάρει θέση για τις ε, διατυπώσεις των τροπολογιών σας. Ε, ένα μόνο ήδη προβλέπετε, μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η ακρόαση στις 27 ε, Φεβρουαρίου το πρωί μέχρι τις 11 και έτσι περνώ στις ψηφοφορίες παραδίδοντας όμως το μικρόφωνο στον πρόεδρό μας, ο οποίος στο μεταξύ έχει καταφτάσει, αλλά φαίνεται ότι έχει εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις. Διακόπτω λοιπόν για λίγα λεπτά. So, colleagues, we Πέντε λεπτά διάλειμμα, αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι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

Συνάδελφοι, σας το να καθίσετε και να βάλετε τις ε, κάρτες ε, στα μηχανήματα για την ψηφοφορία για να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν η δοκιμαστική ψηφοφορία. still two colleagues to vote. We have two colleagues which have put. Δύο. Συνάδελφοι έχουν βάλει την κάρτα μέσα στο μηχάνημα, αλλά δεν έχουν ψηφίσει ακόμα, οπότε του ζητάω να ψηφίσουν και εκείνοι για να ολοκληρώσουμε τη δοκιμαστή ψηφοφορία. Ψηφίστε λοιπόν όλοι. Ε, μία ψήφο ακόμα, ένα συνάδελφο μα λείπει ακόμα. Καλώ τώρα. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις εκθέσεις, την οποία θα ψηφίσουμε σήμερα, ε, του κ. Φων Βατσέκερ και Σμούνιμπον σε ό,τι αφορά την ε, ανάκαμψη και την εξηγήση και του αλούμινου. Ξεκινάμε με την 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ,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 εγκρίνεται συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική E Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα με την, το κατάλογο ψηφοφορία. Λέει ο πρόεδρο, πρέπει να περάσουμε στην. Η συμβαστική τοπολογία ή υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 2,95 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε την τοπολογία 295, άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 301. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 302. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 302. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική K. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 354, όχι, 354 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική NA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 362 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 363 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 364 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 391 υπέρ κατά θα σε ελέγξουμε 391, άρχιτη ψηφοφορία. Μία ψήφος παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 398 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 300 118 συγγνώμη εγκρίνεται 404 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 405 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 407 υπέρ κατά αποχές απο, εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 408 υπέρ κατά ελέγχουμε την το Τροπολογία 408 άρχεται η ψηφοφορία. Ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 409 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε το 409 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 410 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. 124 υπέρ. 124. Όχι, 410 κατέριψε λόγω της 123. Καλώς. 124 υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. 411 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε τη 411. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 412 υπέρ α όχι καταπίπτει. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 413 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 413 άρχη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 414 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 415 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 416 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική R υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 433 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 434 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 435 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 436 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 437 υπέρ, κατά, αποχές Ελέγχουμε την 437 άρχη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Νόμιζα από τους όλοι και ήταν υπέρ. Κάνα λάθος. 438 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 439 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 440 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 441 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 442 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ Α, ναι. Μαζί με την 154 και την 155 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 475 και 76 και 77. Α, όχι, καταπίπτουν. Οπότε περνάμε στην 478 υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, ας ελέγξουμε την 478. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 481 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 482 υπέρ, κατά, ελέγχονται 482, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 483 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε 483. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε τη 484, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. 493 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 494 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 495 υπέρ κατά 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 498 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 500 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 500 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 501 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 502 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 503 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 504 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 504 άρχιτη ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 505 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 520 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 523 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 523, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 524 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 1,72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1,73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5,28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5,29 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Έληξε. Απορρίπτεται. 1,74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1,75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ζήτα συμβιβασμός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5,31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1.76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1.77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.35 υπέρ κατά απορρίπτεται νομίζω ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε αρχίζει ψηφοφορία Λίγη. Απορρίπτεται. 1,78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5,37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1,79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5,38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5,39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.41 και 5.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.43 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε την 543 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μία παραπάνω. 544 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.44 θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία 5.44 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας λήξη απορρίπτεται 5.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στο συμβιβαστικό α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 551 και 552 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 553 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 554 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 555 υπέρ κατά ποχές πρέπει να ελέγξω ηλεκτρονικά λοιπόν την 555 περίεργη κατάσταση Κάποιος δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Λίγη. Εγκρίνεται. από τη 184 μέχρι την 193 μαζί όλες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβιβασμός ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 583 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2-3-2-4 σε μπλοκ εγκρίνεται 2-0-5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2-0-6-2-0-7 εν μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβιβασμός ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2-1-1-2-2 εν μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 2-1-3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνονται από το 592 μέχρι το 596 εν μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο συμβασμός AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AD Συμβιβασμός AD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2, για να το ελέγξουμε, τη 2.20 υπέρ, ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρος, Απορρίπτεται. 2.21 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.22 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά Για το 2022 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψηφό. 223 υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ, δεν το είδα το ΕΛΚ, υπέρ. Λοιπόν, για το 223 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικά παρακαλώ τη 24. άρχεται. Πέρας απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και πάλι ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική αε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική αε α μικρό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AF, ε, συμβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.34 υπέρ κατά τροπολογία κατά, αποχές εγκρίνεται 2.35 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 2.35 ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας πέρας ψηφοφορίας είπα απορρίπτεται 2.36 υπέρ, κατά. Έλεγχος και για τη 2.36 ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.37 υπέρ, κατά. Είστε υπέρ λοιπόν. Είστε κατά. Απορρίπτεται. 2.38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστικός AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.47 υπέρ κατά ηλεκτρονικά 2.47 άρχεται η ψηφοφορία 2.47 πέρας εγκρίνεται 2.48 υπέρ καταπίπτει Ναι. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στη 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AJ συμβιβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ κατά ηλεκτρονικά 255 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.59 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά τη 2.59 άρχεται πέρας εγκρίνεται 2.60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά εγκρίνεται ηλεκτρονικά 261 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 262 και 263 μαζί υπέρ κατά αποχές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 απορρίπτεται. Τώρα για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική πληροφορία άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Πέρας. 49 υπέρ, 3 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια. Vote uh, on uh, και ψηφοφορία για τις διοργανικές συνομιλίες, σύνθεση της ομάδας, όλα αυτά τα γνωστά και δεδομένα, ονομαστικά. Αρχίζουμε. Γιάκοπ, να ψηφίσεις. 50 υπέρ. 3 κατά, 5 αποχές και συγχαρητήρια στους συνεισηγητές. Ελπίζω και στη συνέχεια να έχετε την ίδια επιτυχία. Ίσως και δικιά μου. Now we can move to uh, the GNI regulation report. Έκθεση για τον κανονισμό ε, GNI, ΑΕΠ, τιμές αγοράς. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική D, δέλτα. Α, και πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα τυπογραφικό Αντί για natural, διαβάστε national παρακαλώ, συμβαστική δέλτα υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπερ αποχές εγκρίνεται. 13 υπερκατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται 14, 40 υπέρ κατά αποχές 40 και πάμε στα 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ επαληθεύουμε 46. 46. Πέρας. Και εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20, η συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 7 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ υπερκατά αποχές εγκρίνεται ε, περίφθη 32 υπέρκατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ονομαστικά το σύνολο όπως τροποποιήθηκε αρχίζουμε πέρας Εγκρίνεται λοιπόν με τέσσερι ψήφου κατά και καμία εποχή και τη ψηφοφορία τώρα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αρχίζουμε ονομαστικά πάλι. Πέρας 52 υπέρ, 4 ε, κατά μία αποχή αυτή τη φορά. στο θέμα της ε, ε, έγερσης, μη έγερσης μάλλον αντιρρήσεων για την κατεξοδότηση πράξη της Επιτροπής της 20 Δεκεμβρίου. IDD, αρχικό κείμενο, παράγραφη πρώτη και δεύτερη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τηλογικές αναφορές υπερ κατά αποχές εγκρίνονται, αιτιολογικές σκέψεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και στο σύνολο το κείμενο ονομαστικά. Πέρασε. 51 υπέρ, 1 κατά, 6 αποχές και εγκρίνεται. σχέδιο σύστασης για μη έγερση αντίρρησης σε σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που τροποποιεί τον κανονισμό 1126-2008 IFRS 9 στο Λογιαν. Παράγραφοι 1 και 2 ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται αιτιολογικές ε, αναφορές όλες μαζί υπερκατά αποχές εγκρίνονται, αιτιολογικές σκέψεις on block υπερκατά αποχές εγκρίνονται, σύνολο ονομαστικά. Αρχίζουμε. Πέρας. 50 υπέρ. 4 κατά 4 αποχές. Και συγχαρητήρια. Εκθέση Εμμανουέλ Μαουρέλ. Η υποχρεωτική και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον χώρο της φορολογίας σε σχέση με διασυνοριακές ε, διευθετήσεις, συμβαστική παριθμών ε, ε, α μάλλον, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 81 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 82 υπέρ κατά απο ελέγχουμε την 82 πέρας εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές Επαλθεύουμε Πέρας. Απερίφθη. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 8 και 88 κατά αποχές εγκρίνονται, συμβαστική C κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε ή υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπερκατάποχες εγκρίνεται. Συμβαστική F υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική G υπερκατάποχες εγκρίνεται. Συμβαστική H υπερκατάποχες αποχές εγκρίνεται. Στην 122 τώρα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά επαληθεύεται πιστεύω αλλά στο επαληθεύσουμε Εγκρίνεται δηλαδή. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική ΆΙΟΤΑ υπερκατάποχες εγκρίνεται συμβαστική J υπερκατάποχες εγκρίνεται 33 υπερκατάποχες εγκρίνεται 34 υπερκατάποχες ε, απερίφθη συμβαστική K υπερκατάποχες εγκρίνεται συμβαστική L λάμδα υπερκατάποχες εγκρίνεται 47 υπερκατά αποχές και επαληθεύουμε 47 παρακαλώ Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική M μη υπερκατά αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπερκατά αποχές απερίφθη, 53 υπερκατά αποχές απερίφθη, 54 υπερκατά αποχές απερίφθη 55 υπερκατά αποχές, απερίφθη 56 υπερκατά αποχές, εγκρίνεται 57 υπερκατά Επαληθεύουμε. Πέρας. Συμβαστική εγκρίνεται η 57, ε, νη λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 61 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 61. Πέρας. Εγκρίνεται 62. Α, όχι, έχει καταπέσει. Πάμε στην 63 λοιπόν. Υπέρ. Κατά επαληθεύουμε την 63. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 65 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά επαληθεύουμε την 69 πέρας και απερίφθη 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 74 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 75 υπέρ κατά αποχές οι είναι υπέρ κατά Αχα. ας επαληθεύσουμε λοιπόν Πέρας. Και εγκρίνατε. 76 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε την 76. Πέρας. Εγκρίνεται στην πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε παρακαλώ ονομαστικά. Αρχιτή πέρας 50 υπέρ 2 κατά πέντε αποχές ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα αιτιολογική αναφορά υπερθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έτσι το νομοθετικό ψήφισμα θεωρείται ότι εγκρίθηκε ως τροποποιήθηκε και συγχαρητήρια στον εισηγητή. σύσταση για σύμφωνη γνώμη στην διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για προληπτικά μέτρα στην ασφάλιση και αντασφάλιση. Ψηφίζουμε τη σύμφωνη γνώμη ονομαστικά αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Παίρνετε υπέρ, δύο κατά, έξι εποχές και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στους πραγματευτές κυρίως. Τριάντα δευτερόλεπτα διάλειμμα. Uh, Και ψηφίζουμε την έκθεση Zander Loans, Τραπεζική Ένωση, τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 89 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 92 υπέρ κατά αποχές Απερίφθεια νομίζω, αλλά ας το 92. Πέρας. Και απερίφθη 90 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική α υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 101 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 103 υπερκατά κατά αποχές απερίφθη συμβαστική B υπερκατά αποχές εγκρίνεται C υπερκατά αποχές εγκρίνεται D υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται E ε υπέρ αποχές εγκρίνεται 114 υπερκατά αποχές απερίφθη 124 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 125 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 126 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 117 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 119 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές ε, απερίφθη συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε παρακαλώ 146 Πέρας. Και εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά 150 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, H συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική I, J, προφορική τροπολογία, πράσινη. Ο εισηγητής πρώτα. Ε, ναι, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ όλους σας και για την ευκαιρία να γίνει η ψηφοφορία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάστηκε επιπλέον χρόνος Θυμάμαι πολύ καλά ότι είχατε πει πω ε, εάν χρειαστό θα δίνονταν και παράταση, δεν χρειάστηκε όμω και ευχαριστώ. Θέλω να προβάλλω αντίρρηση στην προφορική τροπολογία γιατί αντίκειται στο πνεύμα, το πολύ επικοδομητικό πνεύμα με το οποίο έγιναν οι συνομιλίε μα με, με τους κοιόδης εισηγητές και γι' αυτό θέλω να προβάλλω αντίρρηση στην προφορική αυτή τροπολογία. Καλώ. ψηφίζουμε την ε, συμβαστική χωρί την προφορική τροπολογία. Ε, πρέπει για λόγους τυπικούς τέσσερις συνάδελφοι από την ομάδα σας έστω να σηκώσω το χέρι καλώς συμβαστική γιώτα χωρίς την προφορική παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και σου οι 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική K K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 212 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική L λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική M μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται π υπερκατά εγκρίνεται συμβαστική Q υπερκατά αποχές εγκρίνεται R υπερκατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 238 υπερκατά αποχές εγκρίνεται 242 υπερκατά αποχές και επαληθεύουμε Πέρας. Απερίφθη. Με μία ψήφο διαφορά. 255 υπέρ κατά. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. S συμβαστική υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 245 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απερίφθη 267 υπερκατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική ταφ τι υπέρ με μια προφορική ο εισηγητής. Το ίδιο ισχύει και για αυτήν εδώ πρόεδρε με το ίδιο σκεπτικό. Για να δούμε χέρια όμως. Καλώς. Χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 269 προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπάρχει αντίρρηση. Τέσσερα χέρια παρακαλώ χωρίς ε, την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απερίφθη 278 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική U ε, υπέρ κατά αποχές απερίφθη Α, συγγνώμη, εγκρίθηκε. Μισθό συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 287 υπέρ κατά και επαληθεύω. Πέρας. Εγκρίνεται 288 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική X χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Y, δηλαδή α με προφορική τροπολογία του εισηγητού, δηλαδή ουσιαστικά προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ε, είτε απλώ τη το όνομα α ε, λοιπόν υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. 320 υπέρ κατά. Ελέγχουμε την 320, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 327 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 335 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο παράγραφος 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AA αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 386 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται 389 με προφορική τροπολογία Περβάνης παρακαλώ ναι θα ήθελα να προτείνω στον ε, συντάκτη της προφορικής ε, τροπολογίας να την ε, τροποποιήσει και να την διατυπώσει ως εξή. υπάρχουν συνεχιζόμενες συζητήσεις σε ό,τι αφορά την νομική βάση για την δημιουργία του μύθου. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται λοιπόν. 392 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι. 387-88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 390 και 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται το κειμένο σε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σε 3 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οπότε τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αρχικό κείμενο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 9 υπέρ, α όχι κατά πίπτη 9, περνάμε κατευθείαν στην 18. 18 λοιπόν 19 κατέπισε και αυτή, οπότε πάμε στη 18 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία 18. No. Vote is η Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Όχι. Καταπίπτει. Ήρθε. Υπέρ λοιπόν της 7. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. λογική αναφορά 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται citation 8 για τις 8 έως 14 ψηφίζουμε. Όχι, διορθώνει ο Πρόεδρος. 7 έως 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Citation 10 τώρα υπέρ. Ναι, από κοινού λοιπόν. 10 έως 14. Citation 10 έως 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Πρέπει να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε λοιπόν τις 10 έως 14 αιτήσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρινούνται. 12. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σατέσιον 16 έως 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά να ελέγξουμε. Τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν 14 υπέρ, Κάνει λάθο ο πρόεδρο. Ήδη ψηφίσαμε τι 14. 15 λοιπόν υπέρ, κατά εποχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά εποχέ εγκρίνεται. Citations 26 και 27 από κοινού υπέρ, κατά εποχέ εγκρίνονται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά εποχέ εγκρίνεται, citations 28 και 29 από κοινού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, citations 30 έως 33 από κοινού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται, τροπολογία 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, citations 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 22 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 27 καταπίπτει οπότε περνάμε στην 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 30 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Περνάμε στην 79 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται, απορρίπτεται, συγγνώμη, 32 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται, 67 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται, 33 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται, ε, συμβαστική ID υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται, συμβαστική 43 ε, υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε τροπολογία 43, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική AFE υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική AG υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 69 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την τροπολογία 82 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στο σύνολο. Στην ε, ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία έτσι όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας, στη ψηφοφορία 48 ψήφοι υπέρ 7 κατά και 2 αποχές ε, τα συγχαρητήριά μας στον εισηγητή και σε όλη την ομάδα του Πάμε στην ε, σχέδιο έκθεση του Λουίτζι Μόργανο σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του συστήματο τη Ευρωπαϊκής Ένωση των Ιδίων Πόρων. Συμβαστική A, B, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική A, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχέ, ελέγχουμε την τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Συμβαστική B υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Με την μαγική ψηφοφορία. Α, όχι. Έχουμε μια προηγούμενη έκδοση του καταλόγου ψηφοφορία, λέει ο So, 29 in 29 υπέρ. Κατά. Τροπολογία 29 λοιπόν, έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στον ε, κατάλογο ψηφοφορίας των σοσιαλιστών. Υπέρ λοιπόν, της 29. Κατά. Ελέγχουμε λοιπόν τροπολογία 29 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην 28 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά ελέγχουμε την τροπολογία 31 πέρας εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την τροπολογία 33 νομίζω πως απορρίπτεται αλλά για να δούμε Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική E υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ, κατά, ελέγχουμε τροπολογία 91. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική A, A μικρό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και ονομαστική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 39 ψήφοι υπέρ, 13 κατά και 3 αποχές. Τα συγχαρητήριά μας στον εισηγητή. Okay. Λοιπόν, και έχουμε και μία ακόμα σελίδα που είναι με συγχωρείτε. Συνάδελφοι, συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε και τώρα μια ψηφοφορία για τον διορισμό του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Γνωμοδοτική Επιτροπή. Μία υποψηφιότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπότε αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, νομίζω ότι διαβοής. Πολύ ωραία. Μαρτουτσέλο. Συγχαρητήρια. Αγαπητέ κύριε Μαρτουτσέλο, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και μπορούμε τώρα να κλείσουμε το εντατικό αυτό κομμάτι που ήταν η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης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 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακαλέσω όσους θα συμμετέχουν στο επόμενο κομμάτι της ημερήσιας διάστατης που είναι το σεμινάριο για τον ανταγωνισμό να παραμείνουν στην αίθουσα και τους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν εδώ αμέσως για να ξεκινήσουμε μια και έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα ήθελα λοιπόν... Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να συζητήσετε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών ή οτιδήποτε άλλο, αν το κάνετε εκτός εθούσης θα μας διευκολύνετε. Για να ξεκινήσουμε τώρα με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι μία συνάντηση της ομάδας εργασίας για θέματα ανταγωνισμού στο πολύ σημαντικό θέμα που είναι ο ανταγωνισμός στις αερομεταφορές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω όλους εσάς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που έχω τη δυνατότητα να καλωσορίσω εδώ τους ομιλητές μας, που έχουν ήδη φτάσει, αλλά καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω και τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ντουζά είναι εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν με έχουν πληροφορήσει σωστά. Είστε εδώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είστε εδώ. Να είστε. Ο κύριος Ντεμπρόκε και η κυρία Μανταμίωβα, οι οποίοι στην ε, DG Trans και Mobility ασχολούνται με τα θέματα της αερομεταφορές, όπως επίσης στην DG Competition. Σας καλωσορίζουμε και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ για οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει κατά τη συζήτηση. Θα γίνει και... Θα... θα συνταχθεί και ένα έγγραφο το οποίο θα συμπεριλάβει όλες τις διαφάνειες από τις παρουσιάσεις και δύο σημειώματα ε, ενημερωτικά από τους εμπειρογνώμονες και το κείμενο αυτό θα λάβει την οριστική του μορφή αφού τα πούμε σήμερα. Πρέπει να πω επίσης πως δυστυχώς δεν έχουμε εκπροσώπηση από τον ΙΚΑΟ. Θα στείλουν όμως μια γραπτή δήλωση που θα συμπεριληφθεί στην τελική μορφή του εγγράφου που θα καταθέσουμε. Και όπως πάντοτε θα ξεκινήσουμε με την εισαγωγή από τους δύο μιλητές που έχουμε καλέσει. Μεγάλη χαρά για μένα να καλωσορίσω τον κύριο Καϊμίτους που είναι καθηγητής για τα ε, οικονομικά δικτύων από το Ινστιτούτο για την Οικονομική Πολιτική και Έρευνα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της ε, Καρσουρής. Σας καλωσορίζω λοιπόν και στα γερμανικά και τον Παύλο Μέντες Τελεών που είναι καθηγητής για δίκαιο ε, εναέριο και διεθνικό δίκαιο και διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου για το σχετικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Λάιντεν στις κατοχώρες. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω πως θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με τις παρουσιάσεις, δεν θα σας καθυστερήσω, 10 λεπτά ο καθένας. Και ελπίζω να το ξέρετε και με τη σειρά που σας παρουσίασα, ο κύριος Κάι Μήτους θα πάρει το λόγο. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Νομίζω πως οι διαφάνειές μου θα ανέβουν στην οθόνη συντομότατα. Η συζήτηση αυτή θα γίνει όλη στα αγγλικά. Έχουμε και σχεδόν σε όλες τις γλώσσες γερμηνία και σας επιτρέπετε να μιλήσετε και γερμανικά αν επιθυμείτε τώρα αγγλικά, γαλλικά, ό,τι, ό,τι προτιμάτε. Για να ξεκινήσω λοιπόν. Ίσως κάποιοι από εσά θυμόσαστε τις τέσσερις ασιατικές τίγρεις, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κόνγκ, την Νότιο Κορέα και την Ταϊβάν. Τη δεκαετία του 80 που είχαν στοχευμένες στρατηγικές για να κατακτήσουν τις αγορές του κόσμου σε κάποιους συγκεκριμένους κλάδους. Δηλαδή ήταν τα ηλεκτρονικά, τα ναυπηγεία, ο χάλιβας και αυτό δημιούργησε πολύ ε, ανάμεικτα συναισθήματα στις ε, αναπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν κάποια εμπορικά ζητήματα, κάποια αντίμετρα, αλλά τελικά οι χώρες αυτές πέτυχαν. Και τράβηξαν προς τα βρός και την Κίνα, μεγάλη χώρα, και νομίζω σήμερα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε αυτό το μηχανισμό, το, αυτή τη μηχανή ανάπτυξης ε, στην Ανατολική Ασία. Μιλάμε τώρα για τις χώρες του κόλπου, τα Εμμυράτα και το Κατάρ, που προσπαθούν να γίνουν αντιστοίχω τίγρης και δεν στοχεύουν στην αγορά των ηλεκτρονικών, αλλά στις υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα ε, στις μεταφορές. Και εδώ θα συμπεριλάβουμε και τις διεθνείς αερογραμμές. Ίσως λοιπόν θα αποτελέσουν τον κλάδο που θα αναπτύσσεται στο μέλλον και να σας πω πως και εδώ έχουμε τέτοιου είδους ε, συγκρούσεις και έχουμε και μια άλλη ομάδα που είναι οι αναδυόμενες μεγάλες αγοράς όπως η Κίνα, η Τουρκία και οι χώρες αυτές έχουν μια τεράστια ε, εγχώρια αγορά σε αντίθεση με τις μικρές χώρες ε, όπως το Κατάρ και τα Εμμυράτα και που θέλουν επίσης να μπουν στην αγορά των αερογραμμών αλλά δεν θέλουν να ανοίξουν ε, τις δικές τους εγχώριες αγορές υπερβολικά στον ε, ανταγωνισμό. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ποια είναι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε να έχουμε σταθερή οικονομική ανάπτυξη, σφρεγγυλή ανάπτυξη χώρες αυτές και να ενταχθούν στην παγκόσμια οικονομία και βεβαίως θα πρέπει να ακολουθούν δίκαιες πρακτικές και να μην ε, παρεμβαίνουν υπερβολικά κυβερνήσεις. Αλλά για κάποιο διάστημα ακόμα νομίζω θα πρέπει να μπορούμε να δεχτούμε ότι σε κάποιο βαθμό θα έχουν κάποιες επιλεκτικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Τώρα, ακούγονται πολλά. Δηλαδή, ότι οι αερογραμμές επιδοτούνται με διάφορους τρόπους, δεν έχουμε πάντα τους αριθμούς, αλλά επιπλέον ε, μιλούν πολύ συχνά όσοι τους καταγγέλουν για διαφάνεια, Γιατί έχουμε εδώ πέρα και χρηματοδοτικά μέσα κρατικά και αεροδρόμια κρατικά και αερογραμμές κρατικές, οπότε κανείς δεν μπορεί να δει αν κυκλοφορούν επιδοτήσεις. Οπότε ε, έχουν και την έλλειψη ανοίγματο των εγχωρίων αγορών και οι βασικές αρχές για την για το δίκαιο εμπόριο είναι καταρχήν ΠΟΕ και ΓΚΑΤΣ που δεν ε, ισχύουν για τις αερογραμμές γιατί εκεί έχουν το δικό τους καθεστώς για τις αερομεταφορές που δεν αναφέρεται καθόλου στα εμπορικά θέματα. Μπορούμε βεβαίως να μιλήσουμε για τις αρχές του ΠΟΕ. για τις ενισχύσεις, για τα αντίμετρα, τα τις ενισχύσεις που δεν επιτρέπονται και για τους δασμούς ως αντίμετρα μπορούν να επιβληθούν. Αυτοί λοιπόν οι θεσμοί αντίμετροι για να επιβληθούν πρέπει να τεκμηριώνονται με το γεγονός πως υπάρχει ενίσχυση, βλάβη και σχέση άμεση μεταξύ ενίσχυσης που καταβάλλεται και βλάβης που έχει τυπωστεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το κριτήριο αυτό και να σας πω πως όντως υπάρχουν κάποιες αρχές στις όλοι ακολουθούν, αλλά οικονομικά, να σας πω πως τα αντίμετρα πολλές φορές ε, στηρίζονται πρώτος στο γεγονός ότι τις χώρες που εισάγουν αυτές τις πληροφορίες τις προστατεύουν από στρεβλώσεις, από υπερβολικό κόστος και βεβαίως είναι διορθωτικά μέτρα για τη χώρα που εξάγει αυτές τις υπηρεσίες μια και τους επιτρέπει να καταλάβουν πως δεν μπορεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική να βασίζεται σε ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Αυτά τα αντίμετρα λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις είναι ε, επικοδομητικά και εδώ έχω... Ποια είναι η λέξη κλειδί. Να είναι κανείς προσεκτικός η σύνεση, γιατί μιλάμε για μεταφορές. Και ο κλάδος αυτός είναι πολύ διαφορετικός από άλλους οικονομικούς κλάδους, γιατί δεν είναι τόσο συνήθιστο να έχουμε εδώ επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις. Γιατί τα αεροδρόμια, για παράδειγμα, αν χρηματοδοτούνται, αυτό είναι συνηθισμένο παντού στον κόσμο. Δεύτερον, αν μιλάμε για αντίμετρα, υπάρχει αμοιβαιότητα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά γίνονται. Για παράδειγμα, Έχουμε τα σλότ στα αεροδρόμια και τις ρήτρε ε, σταδιακής κατάργησης, το grandfathering clause δηλαδή, και είναι πολύ δύσκολο για έναν ανταγωνιστή να μπει σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο και να πάρει σλότ για απογειώσεις προσγειώσεις. Άρα λοιπόν και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν κάνει κανείς μια ευρύτερη αξιολόγηση. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω πως είναι βέβαια ο ανταγωνισμό σε αερομεταφορέ πολύ καλό για τον καταναλωτή, γιατί οι αερογραμμέ είναι ο κλάδο στον οποίο ο ανταγωνισμό καλύτερα λειτουργήσε στο παρελθόν. Και πρόσφατα είχαμε ε, την Air Berlin και την Alitalia που συγχωνεύονται, εν πάση περιπτώσει ενώνονται και έχουν σχεδόν εξαφανιστεί και οι δύο. Και τι ε, σημαίνει αυτό, είναι ε, υψηλότερες τιμές, άρα λοιπόν λιγότερος ανταγωνισμός υψηλότερα κέρδη για τις μεγάλες πέντε αεροπορικές εταιρείες ομίλους, ε, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε την ένταση του ε, ανταγωνισμού και όχι το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από εξωτερικούς ανταγωνισμούς. Και αυτό το λέω ως ε, σχόλιο. Στη σύνοψη να σας πω πως εάν είναι ε, τεράστια και συστηματική η αλλοδαπή αυτή κρατική ενίσχυση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να γίνονται διεθνεί διαβουλευσει και ίσως η απειλή και μόνο των αντιμέτρων να είναι αρκετή. Θα πρέπει όμως να κάνουμε και μια αξιολόγηση τη πρακτική που ακολουθούν οι ξένες χώρες και να δούμε αν πριν αποφασίσουμε ε, αντίμετρα έχουμε λάβει δόντως υπόψη τα τι κάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες γιατί και εμείς επιδοτούμε τα δικά μας ε, αεροδρόμια και οι δικές μας αερογραμμές, αεροπορικές εταιρείες ε, ενισχύονται από αυτό και έχουμε και τα grandfathering ε, δικαιώματα για τα slot οπότε ίσως υπάρχουν αρκετά αντίμετρα ήδη που να ισχύουν και να μην χρειάζονται άλλα η αμοιβαιότητα είναι σημαντική Όποια πολιτική και να επιλεγεί θα πρέπει να μετρηθεί προσεκτικά και με μια ευρεία κατανόηση του ανθρώπινου συμφέροντος. Και το λέω αυτό γιατί στον κανονισμό εμφανίζεται τρεις φορές το human interest, ανθρώπινο συμφέρον. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πει ότι δεν θα λάβουμε αντίμετρα γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποια είναι ο θεμητός ανταγωνισμός, αλλά και αρκετός ανταγωνισμός. Θέλουμε να έχουμε ανταγωνιστές εδώ. Και ίσως θέλουμε να αναπτυχθούν και οι χώρες αυτές. Νομίζω και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα προκύψει όταν ο κανονισμός θα εφαρμοστεί οπότε πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει τον κανονισμό αυτό και όπως είπα σύνεση. Μην είστε υπερβολικά αυστηροί. δεν είναι μόνο οι αερογραμμέ που έχουν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ω πανεπιστημιακό, θα έλεγα πω στον κανονισμό αυτό θα έπρεπε να τον εφαρμόσουμε με επιστημονική αξιολόγηση συλλέγοντα στοιχεία τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο κοινό έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται, να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται και ίσως να καταλήξουμε και σε κάποια διδάγματα τα οποία ε, θα εφαρμοστούν και σε άλλους κλάδους. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ. Εγώ που τήρησα το χρόνο σας. Επακριβέστατα, 10 λεπτά και 0 δευτερόλεπτα. Ο Παύλο Μέντες Τελεών, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, με τον συνάδελφο δίπλα μου εδώ βέβαια, στον οποίο και είναι μεγάλη η χαρά ε, που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα την, ε, τις προτάσεις μου, τις ιδέες μου για το διεθνή ανταγωνισμό στην ε, αεροπορία. Έχω μερικές διαφάνειες και ξεκινώ με την πρώτη όπου διατυπώνω το ερώτημα τι θεωρούμε θεμητό ανταγωνισμό ερώτημα που ίσως να μην απαντούν μόνο οι νομικοί. Η συνθήκη όμως για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην οποία στηρίζεται και η δουλειά μας αναφέρεται σε ελεύθερο ανταγωνισμό και βλέπω σε άλλες οδηγίες γνήσιο ή καθαρό ανταγωνισμό. Αλλού σε άλλα νομοθετικά κείμενα γίνεται λόγος για θεμητό ανταγωνισμό. Τι ακριβώς λοιπόν εννοούμε. Και όπως είπα δεν είναι μόνο νομικό το ερώτημα ε, συνδέεται και με τόσο είπε ο καθηγητής Μήτους μόλις τώρα ο συνάδελφος εάν δηλαδή θεωρούμε πως ε, η συνεννόηση μεταξύ επιχειρήσεων και οι κατάχρηστες πόσες θέσεις είναι ε, αθέμητος ανταγωνισμός ή μήπως και άλλες τε, αντίστοιχες συμπεριφορές. Εδώ πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη βάση, δηλαδή το σχέδιο του κανονισμού κυρίες και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη ένωμη τάξη η οποία περιορίζει τις επιδοτήσεις οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ίνδοι, οι Άραβικές χώρες δεν ρυθμίζουν, δεν περιορίζουν τις επιδοτήσεις. Καλά καλά δεν έχουν αρχίσει να μιλάνε για ανταγωνισμό βέβαια στην νομοθεσία τους. Επομένως, δεν καλύπτεται στον όρο του ε, του ανταγωνισμού η έννοια της επιδότησης στη νομοθεσία των άλλων αυτών νομών τάξεων. Αυτό πρέπει να το ορίσουμε ως πρώτο ζήτημα και αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια παρατήρηση για τον ΠΟΕ και την εφαρμογή τη δυνατότητα καλύτερη εφαρμογής αυτού στις αερομεταφορές Τίθεσε ε, αμφισβήτησα. Γιατί λοιπόν δεν ήταν αποτελεσματικός ο καρονισμός και βλέπω αντίστοιχε παρατηρήσεις και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχέδιο καρονισμού ήταν μάλλον ενδοσκοπική. Βεβαίως θα πρέπει να κοιτάξουμε όλο το τομέα των μεταφορών, τις βασικές αρχές της Σύμβασης του Σικάγο, άλλες συμφωνίες διεθνείς και ούτω καθεξής. Ωστόσο ο κανονισμός εξέει δεν μπόρεσε να εφαρμοθεί επειδή υπάρχει το καθεστώς του Σικάγο που προσδιορίζει η Σύμβαση του Σικάγο σε πρώτο λόγο και οι λοιπές ε, συμφωνίες. Η Σύμβαση του Σικάγο λοιπόν δεν μιλάει για θεμητό ανταγωνισμό, επιτρέπει στα κράτη τον προσδορισμό των παρεχομένων υπηρεσιών και για να περάσω στην επόμενη διαφάνεια έχει κλειστούς εναέριους χώρους ορίσει αυτή η ε, σύμβαση. Για διάφορους λόγους δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Κλείνουμε τον αέριο μας χώρο, τον ανοίγουμε μόνο σε ε, εκείνους που ικανοποιούν τους όρους. Ωστόσο, οι συμφωνίε για παροχή αεροπορικών υπηρεσιών δεν μιλούν απαραίτητα για συμφωνία. Ούτω ή άλλω δεν είναι πολύ ευνοϊκέ στον ανταγωνισμό, γιατί έχουν ε, συχνά διατάξει οι οποίε αντίκειται στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Επομένω, τίθεται το ερώτημα του συνδυασμού ή της ε, συμφιλίωσης του περιορισμένου, της περιορισμένης παροχής ε, με προκαθορισμένες συμφωνίες, συμφωνίες αερομεταφορών αυτών των υπηρεσιών με τις αρχές για τον ε, ελεύθερο ανταγωνισμό της συνθήκης για τη λειτουργία και την ελεύθερη δυνατότητα των ελεύθερων ταγωνιστημών. Ο κύριος Μήτους μας λέει ότι είναι απαραίτητη η αμοιβαιότητα. Έστω ναι, συμφωνώ, πρέπει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να συγκεράσουμε τις διαφορετικές θέσεις. Το πώς θα γίνει βέβαια είναι μεγάλη πρόκληση. Και εκεί που λέω στην ε, τρίτη τελεία, οι αεροπορικές εταιρείε μερικές φορές είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται ακόμα και αντίθετα με όρους ε, ε, ανταγωνισμού ε, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερο δυναμικό. Και άλλωστε το ξέρει αυτό η Επιτροπή, γι' αυτό υπάρχουν διαφορές υποθέσεις που εξετάζει η Επιτροπή με την υποψία του καρτέλ και παραπέμπει αντιστοίχως στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο ελέγχουν οι κυβερνήσεις. Ε, θέλουμε, το είπε και ο κύριος Μητούς, να μπορούν οι κρατικές αρχές να ελέγχουν και βέβαια και οι αρχές ε, πολιτικής αεροπορίας και να ελέγχουν αυτές τις εργασία, να ε, ενισχύουν βεβαίως και για άλλους λόγους, να ενισχύουν και την συνδεσιμότητα, τους ε, διαφορετικούς προορισμούς κτλ. Και για να περάσω στην επόμενη διαφάνεια, ενώ ο προτινόμενος κανονισμός προσανατολίζεται όπως είναι κατανοητό ε, στην υλοποίηση των αρχών της ελεύθερης αγοράς που έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός παραμένει για μένα το ερώτημα και σε αυτό επίσης τοποθετήθηκε ο συνάδελφος νωρίτερα. Παραμένει λοιπόν για μένα το ζήτημα της πρακτικής εφαρμογής των διατάξεων του, γιατί αυτό ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί. Δεν ξέρουμε πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη. Πώς μπορεί η Επιτροπή δηλαδή σε μια συμφωνία της οποίας δεν είναι μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνει στη χώρα, Φερρυπίν την Ινδία και να πει άθελο να μου πεις τι είδου συμφωνίε έχεις». Θα πάει να χτυπήσει την πόρτα στον η Επιτροπή να πει «Θέλω δηλώσεις, ε, οικονομικά δελτία και ούτω καθεξής». Εγώ λοιπόν προτείνω μία λύση που μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμα, χρήσιμη. Τι είναι η αεροπορική εταιρεία. Δεν το ορίζεται, ορίζεται μόνο στην ε, σύμβαση του Σικάγου. Εντάξει, το ξέρω αυτό στον κανονισμό 1028 επίσης εξαιρετικός κανονισμός, καταπληκτική διατύπωση που μας λέει ότι είναι μια επιχείρηση η αεροπορική εταιρεία. Πολύ ωραία, συμφωνώ. Φρονώ ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συνομιλεί με τρίτες χώρες πρέπει να τους λέει οι εταιρείε σας, οι, οι αεροπορικές, ε, οι αερομεταφορείς σας μάλλον, οι οποίοι αναλαμβάνουν μεταφορά προσώπων από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι επιχειρήσεις και να έχουν αντίστοιχα να πληρούν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις ε, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει βέβαια η θεωρία η νομική που έχουν υιοθετήσει πολλά δικαιοδοτικά όργανα ε, στον κόσμο σε σχέση με τις κρατικές επιδοτήσεις για το πού μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Αρχή η αντίστοιχη να αναλάβει δράση σε περίπτωση παρέμβασης μίας επιχείρησης που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εσωτερική αγορά ε, κατά τρόπον ώστε να την διαταράσει και αυτό το ανέφερε και ο καθηγητής Μήτους και η ΚΑΟ βέβαια έχει αντίστοιχα προτείνει λύσεις. Ε, με μία απόπειρα ο θεμητός ανταγωνισμός να περιγραφεί ως βασική αρχή, το λέω έτσι με πολύ επιφυλακτικό τρόπο, χωρίς όμως να μπορεί να δεσμεύει ακριβώς τα μέλη της, τα συμβαλόμενα της ε, μέρη ή καο στον προσδορισμό αυτής της αρχής. Σας ευχαριστώ θερμά, ολοκλήρωσα εδώ τις διαφανίες μου και είμαι στη διάθεσή σας για την περαιτέρω συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε και τον χρόνο σας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βέβαια έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να προβούμε σε συζήτηση. Συνάδελφοι, ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ποιο από τους δύο τους ελεύθερου θα πάρει το λόγο. Ναι, μόνο δύο από εμά ενδιαφερόμαστε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε ε, πολύ για αυτές τις παρουσιάσει. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα γιατί ο πρώτος ομιλητή ανέφερε ότι εδώ οι επιχειρήσεις ε, της, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υγιείς. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρκούντος υγιείς ε, σε σύγκριση με τα όσα μας περιμένουν. Δηλαδή υπάρχουν τώρα αερομεταφορείς ε, από τις χώρες του κόλπου αλλά και άλλες αερομεταφορείς ε, με, με πολλά χρήματα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν εδώ σε μια αγορά δηλαδή με δυνητικά 500 εκατομμύρια επιβάτες. Και ταυτόχρονα ζητούμε από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναδιαρθρωθούν. Ε, θεωρείτε πως είναι θεμητό να ζητούμε να υπάρχει ε, οικονομική ε, διαφάνεια στο πλαίσιο των ε, μελλοντικών συμφωνιών που θα συνάψουμε στο επίπεδο των αεροπορικών μεταφορών. Γιατί και εσείς ο ίδιος είπατε ότι αν τέτοιου είδους ενισχύσεις εφαρμόζονται μονίμως, τότε ενδεχομένως να πρέπει να αναλυφθεί δράση. Και η οι αερομεταφορείς Ευρωπαίοι εκφράζουν αυτές τις ανησυχίες. Δηλαδή αν δεν αλλάξει κάτι και οι εν λόγω επιχειρήσεις της αεροδαπής δηλαδή εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να αλλάξει τίποτα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, και κάτι ακόμα ε, ενημερωτικά εδώ προς το κοινό. Η Air France, η British Airways και η Lufthansa ε, έχουν καθεμία 10 με 12 Airbus 380. Ε, ενώ η Emirates έχει 350. Airbus 380 πάντα. Άρα λοιπόν, Λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα προσωπικά στοιχεία που έχουν τέτοιου είδου επιχειρήσει. τι είδου μοχλό για την άσκηση πιέσεων διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κάτι δική μα άποψη. Ποια είναι η δική σα ε, άποψη, κύριε καθηγητά. Μέσα σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ναι, ε, ακριβώς η διαφάνεια είναι ε, το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι το ιδιαίτερο ε, σε σχέση με τον κανονισμό και ο Στάνθος αναφέρθηκε σε αυτό, δηλαδή το πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερη διαφάνεια τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περισσότερη οικονομική διαφάνεια και αν θα μπορούσε αυτό να είναι ο στόχο, ο βασικό στόχο τη ε, πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει, αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Γιατί ε, θα ωφελήσει τι επιχειρήσει μακροπρόθεσμα. Πραγματικά δηλαδή, ε, εδώ βεβαιώνω τα όσα μόλι μα είπατε. Οι πέντε μεγάλοι μα αεροπορικοί όμιλοι βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση. Δηλαδή η αξία των μετοχών τους ε, δεν είναι αυξανόμενη, οπότε δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, που να αντιμετωπίζουν. Και βέβαια, αν ο κανονισμός εγκριθεί, και θέλει να τον αξιοποιήσει περαιτέρω Επιτροπή. Εγώ τι λέω απλώς, δεν χρειάζεται να βιαστεί, θα πρέπει να αναλογιστεί καλά τα επόμενα βήματα στα οποία θα προβεί. Και θα πρέπει λοιπόν να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα τη διαφάνεια. αξιώνοντα από αυτέ τι υπόλοιπε επιχειρήσει που θα εισέλθουν στην αγορά, να καταδείξουν πώ εξελίχθηκε η οικονομική του κατάσταση, ποια είναι τα βασικά δηλαδή στοιχεία τη οικονομική του κατάσταση, καθώ κάτι τέτοιο θα βοηθούσε. Ο δικό μου φόβο είναι ότι αυτέ οι μεγάλες αεροπορικές ε, ε, θα δηλαδή στήσουν πιέσει προκειμένου να γίνουν περισσότερα βήματα από τη μας πλευρά, ταχύτερα, χωρί ακριβώ να γίνει ε, ε, ο κατάλληλο έλεγχο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο Βόλφκανγκ έχει τώρα το λόγο. Κύριο Κλίντ. Σα ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε, ότι οι κανόνε δηλαδή του ΠΟΕ δεν ισχύουν για τον τομέα των αερομεταφόρων. Δεν θα ήταν χρήσιμο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί θυμάμαι ότι όταν αναφερόμαστε στους ε, κατασκευαστές αεροσκαφών, δηλαδή την Boeing και την Airbus, ε, εκείνοι είχαν ε, δώσει μάχη για πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά τους κανόνες κατά του αθέμητου ανταγωνισμού με βάση ακριβώς το πλαίσιο του ΠΟΕ. Ε, βέβαια τελικά κατάφεραν να φτάσουν σε μια συμφωνία μεταξύ τους αυτοί οι δύο κατασκευαστές, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει αν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα σενάριο στο πλαίσιο του οποίου οι εν λόγω κανόνες του ΠΟΕ δηλαδή θα ίσχυαν και για τους αερομεταφορείς, τότε τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Γιατί νομίζω ότι η πρόταση την οποία κάνατε, ότι θα πρέπει δηλαδή να αξιώσουμε περισσότερη διαφάνεια, με άλλα λόγια να έχουμε περισσότερα, περισσότερη πρόσβαση στους ολογισμούς, στα βιβλία και στοιχεία των ε, ε, λόγω επιχειρήσεων, θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν νομίζω δηλαδή πως οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι Κατάροι, οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, η Emirates, η Etihad, να είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία τους. Και ακόμα ε, και αν το έκαναν, ε, γιατί βέβαια ορισμένες που είναι σημαίνει στο χρηματιστήριο τους άλλους έχουμε κάποια πρόσβαση στα στοιχεία, αλλά ε, ειδικότερα από, σε ό,τι αφορά την Καταρέρ, την Emirates και άλλες, ε, καθώς λαμβάνουν ακόμα κρατικές ενισχύσεις, δεν θα ήταν διατεθειμένες να μας δώσουν πρόσβαση στα κάτω στοιχεία. Ε, και αν το έκαναν ενδεχομένω να μαγείρευαν το εισαγωγικό λίγο τα στοιχεία που θα σα έδιναν. Εντάξει, ίσω λέει, είμαι λίγο υπερβολικό εδώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ε, κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί. Το να λέμε ότι οι δικοί μα ε, αερομεταφορεί βρίσκονται σε καλή, σε υγιή κατάσταση, ναι, ισχύει, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι αερομεταφορεί που είναι, βρίσκονται πρώτη σε εξάλληψη, όπω η Αλιτάλια για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, αυτό που διαπιστώνουμε και εδώ περνάω στο δεύτερο ερώτημά μου, είναι οι αερομεταφορείς χαμηλών, χαμηλού κόστους, οι οποίοι ε, αυξάνονται όλο και περισσότερο. Η Ryanair, ναι, για παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη πλέον από τη Lufthansa. Μετέφερε δηλαδή πέρσι περισσότερους επιβάτες. Άρα, οι μεγάλες απειλές που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το τομέα προέρχονται από τον αθέμητο ανταγωνισμό από άλλους εξωτερικούς αερομεταφορείς ή και από διαφορετικές ε, συνθήκες, συνθήκες δηλαδή στην αγορά οι οποίες ε, δεν τους επιτρέπουν να είναι ανταγωνιστικές και εδώ αναφέρομαι στις μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Lufthansa, η Air και άλλες. Δηλαδή αν δούμε και τις ε, αμοιβές, για παράδειγμα εκεί που ισχύουν, είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που ισχύουν στην EasyJet, η Ryanair και άλλες. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο και τις συνθήκες εργασίας και τις, ε, τις δομές παροχής αυτών των υπηρεσιών στα δύο διαφορετικά είδη επιχειρήσεων. Ποιο θέλει να απαντήσει. Με το μικρόφωνο παρακαλώ. Έχετε δίκιο. Η λειτουργία αυτών των αερωματοφορών δεν επιπτεί στα καθεστώτα GATS και ΠΟΕ για συγκεκριμένους λόγους και η πρότασή σας Δηλαδή, και μιλήσατε για τις διαφορές μεταξύ Airbus και Boeing, αλλά αυτό είναι το προϊόν. Το αεροσκάφος είναι το προϊόν και εμείς μιλάμε εδώ για υπηρεσίες. Και αυτή είναι μια σημαντική διάκριση η οποία πρέπει να γίνεται. Ε, τούτου λεχθέντος νομίζω ότι η ε, υπηρεσίες για παράδειγμα συντήρηση, διανομή κτλ ε, εμπίπτουν στην ε, γάτς για την υπηρεσία αλλά και πάλι για την παρουσίαση που κάνουμε εδώ και τη συζήτηση τα θέματα αυτά δεν είναι σχετικά όπως είπατε και εσείς γιατί να μην εφαρμόσουμε τους κανόνες κατά των κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν, που ισχύουν στον ΠΟΕ και στην ΓΚΑΤΣ για την ε, παροχή υπηρεσιών αερομεταφορών. Είναι μια υγιής πρόταση που θα μπορούσε να γίνει όμως οι αερομεταφορές δεν εμπίπτουν ακριβώς λόγω των εντάσεων που υπάρχουν μεταξύ των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουμε εμείς να, μετα... να ισχύσουν και σε αερομεταφορές και στις τρίτες χώρες που δεν το επιθυμούν. και που ρεαλιστικά, το είπατε και εσείς, δεν θέλουν να ανοίξουν ε, τις χώρες τους και θέλουν οι αριμετοφορές να παραμείνουν ως ε, εργαλείο ε, πολιτικής. Είναι ένα εμπορικό εργαλείο χάραξη πολιτικής και άσκηση πολιτικής και γι' αυτό επιθυμούν να κρατήσουν το θέμα αυτό εκτός των κανόνων για ενισχύσεις, για ανταγωνισμό κτλ και για τις αερογραμμές τους και για τις υπηρεσίες που προφέρουν, για την Κατάρ. Ναι, είναι δύσκολος αντίπαλος. Η Emirates ίσως είναι λίγο πιο ανοιχτή και πιο προσπελάσιμη. Τουλάχιστον αυτό ακούω σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Και υπάρχει μια κάπως ασαφής δομή που κυριαρχεί σε όλες τις αερογραμμές και δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε εμείς να βρούμε. Ίσως εσείς θέλετε να ασχοληθείτε. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση προς την πρώτη ερώτηση. Ναι, είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε με ένα παγκόσμιο ομοιογενές καθεστώς. Ο κανονισμός αυτός όμως έχει σκοπό να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Οπότε ναι, είναι επικοδομητικό στοιχείο αυτό στον κανονισμό και για την αγορά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξιοσημείωτο το ότι οι γνωστοί αερομεταφορείς όπως η Λουσχάντζα είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις. Δεν είναι τόσο πολύ ο αριθμός επιβατών, γιατί οι low cost έχουν περισσότερους επιβάτες πια, αλλά παρόλα αυτά οι άλλες αεροπορικές εταιρείες είναι κερδοφόρες. Ζούμε σε μια εποχή ανάπτυξης και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί όταν θα φτάσει η επόμενη κρίση. Αν όμω συνεχίσουν τα πράγματα όσοι έχουν, τότε νομίζω ότι οι πέντε όμιλοι αυτοί είναι ικανοποιητικοί, δύο μεγάλωσαν, αλλά με πέντε όμιλ, ε, ομίλους που είναι διαφοροποιημένοι, που είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους, που έχουν διαφορετικά μερίδια και εξυπηρετούν. Νομίζω ότι έτσι όπως έχει κατάσταση θα ανησυχούσα περισσότερο για τον ανταγωνισμό και δεν θα ήταν καλό να έχουμε κάτω από πέντε. Και υπάρχουν κάποιες ε, αντιρρήσει, κάποιοι οικονομολόγοι λένε πως δεν είναι αρκετά μεγάλη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίζει πέντε ομίλου τέτοιου μακροπρόθεσμα, οπότε μετά την επόμενη κρίση θεωρούν πως ένας από αυτού να εξαφανιστεί και να τον αγοράσουν οι υπόλοιποι. Αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει κάτι τέτοιο. Αυτό που βλέπουμε είναι ανάπτυξη και οι πέντε είναι επαναλαμβάνουν σε πολύ υγιή κατάσταση. Αλλά για τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στηρίξει πέντε ομίλους, τότε θα έπρεπε να ψάξουμε για μεγαλύτερες περιοχές, για ένα όραμα Ευρωπαϊκή Ένωση συν Μέση Ανατολή. για να έχουμε 5, 6, 7 ομίλους εκεί και σε επίπεδο ανταγωνισμού αυτό είναι και το καλύτερο. Σύντομα παρακαλώ. Μια ακόμη ερώτηση αν μου επιτρέπετε. Εσείς φρονείτε ότι έχουμε θεμητό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ρωτώ διότι Γνωρίζουμε ότι ε, εν γέννη υπάρχει έλεγχος στην πρόσβαση στην αγορά. Δηλαδή δεν υπάρχει μια γνήσια ανοιχτή αγορά των ε, μεταφορών. Χρειάζονται παραδείγματι οι χρονοθυρίδες, τα σλότ. Ιδάλλως δεν μπορεί κανείς να μπει στην αγορά αν δεν εξασφαλίσει σλότ. Άρα δεν υπάρχει θέμα του ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά ακριβώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε είναι αυτό τον σλότ για τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή τον θεμητό ανταγωνισμό. Αλλά υπάρχει προηγούμενο σταδιακής εισαγωγής στη δεκαετία του 90 του θεμητού ανταγωνισμού του ανοιχτού ανταγωνισμού. Χάσαμε δύο αεροπορικέ εταιρείε, έχουμε όμω πέντε μεγάλου ομίλου που φαίνονται βιώσιμοι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον και για το εγγύ μέλλον, για το ορατό μέλλον. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Οι διεθνείς αγορές βέβαια αναπτύσσονται ταχύτατα. Με φορείς που διωγγώνονται διαρκώς και παίρνουν μεγάλο κομμάτι από την πίτα. Αλλά και οι δικές μας εταιρείε μεγαλώνουν επίσης. Ας μην είμαστε υπερβολικά επιθετικοί απέναντι τους. Έχουν 50% της ευρωπαϊκής αγοράς ή ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όμιλοι. Επομένω, νομίζω ότι είναι ε, δίκαιη η κατανομή. Ο κύριος Μέντες Τελεών, ε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση σας. Δεν έχει τεθεί το θέμα τόσο πολύ του ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού, που είναι ένα στοιχείο του ελεύθερου ανταγωνισμού, μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Υπάρχει πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά. Ασφαλώς έχετε δίκιο όταν επισημαίνετε ότι κάποιες, ε, ε κάποιοι αεροπα, ε, αερομεταφορείς μειονεκτούν όταν είναι υποχρεωμένοι να ξεκινούν ε, την, τα δρομολόγια τους από αεροδρόμια που θεωρούνται ακριβά, είναι ακριβά όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο. Ενώ για Α, άλλα αεροδρόμια ίσως δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα χρήσης. βέβαια δεν είναι μόνο, δεν εξατελείται εκεί το, ισότιμο, το πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού ή θεμητού ανταγωνισμού. Γιατί η λειτουργία και παροχή αεροπορικών υπηρεσιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά πολύ ωραία εναρμονισμένη με τον 108 υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που δεν είναι αρμονισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. εργασιακέ εργασιακές σχέσεις, σχέσει. φορολογικές σχέσεις, η Ryanair και μπορεί να μου πείτε ότι είναι και σωστό ή πάντως κατανοητό. Εκμεταλλεύεται αυτές τις διαφορές. Υπάρχουν πολύ ευέλικτες νομοθεσίες, έχουν ε, τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν από το Δουβλίνο το προσωπικό τους με αυτή την ευέλικτη νομοθεσία και αν υπάρχουν ε, διάφορες προσφυγές σε δικαστήρια γιατί προσωπικό που εδρεύει στη Μασαλία πάλι υπάγεται στο Ιρλανδικό δίκαιο. Ε, φορολογικά πλεονεκτήματα επίσης. Όταν ε, το να, το να επιλέξει κανείς έδρα ε, εταιρεία ε, στο Παρίσι ή το Δουβλίνο αλλάζει πάρα πολύ το, το φορολογικό βάρος. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τι εννοούμε ως θεμητό ή ανταγωνισμό. Διότι δεν είναι αρμονισμένα όλα αυτά τα παιδεία πολιτικής. Έτσι είναι η ζωή όμως και ο νόμος. Ο πρόεδρος, αν μου επιτρέπετε, ας ε, κάνω και εγώ μια παρέμβαση, μια ερώτηση. Νομίζω πως ε, περιγράψατε με σωστό τρόπο το γενικότερο περιβάλλον γιατί μπορεί να έχει και πολιτικό χαρακτήρα η απόφασή μα, ε, Δηλαδή στι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, για παράδειγμα, ακριβώ ε, η αγορά έχει πιο πολιτική χρειά, ειδικότερα μετά από την τελευταία οικονομική κρίση. Προσπάθησαν ακριβώ οι Αμερικανοί να, να εξηγιάνουν και πάλι τον γενικότερο τομέα. Που έγινε αυτή η προσπάθεια να διοργάνωση του συνόλου τη αγορά. Άρα λοιπόν, κατά τη δική μου αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμε μια προσέγγιση πιο πολύ προσανατολισμένη στην αγορά. Δηλαδή όταν συμβαίνει κάτι βλέπουμε ακριβώ σε ποιου έχει προκύψει το πρόβλημα και από εκεί και μετά εκείνο που λείπει είναι μια στατική. Δηλαδή λαμβάνοντα υπόψη τα όσα μας περιγράψατε σε ό,τι αφορά την εργασιακή νομοθεσία και ούτω καθεξή, το ζητούμενο είναι να θα αναπτύξουμε ενδεχομένω μια στρατηγική για να δούμε πώ μπορούμε να κατευθύνουμε την αγορά ή να αφήσουμε την αγορά να κατευθυνθεί ανάλογα με το πώ εκείνη θα κατευθυνθεί. Όπω ε, για παράδειγμα συνέβη στην περίπτωση σε Μπερλίν που την αφήσαμε έτσι και τελικά κάποιο βρέθηκε ε, για να αναλάβει εκείνη. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένω να καταλήξουμε ε, στην κατάσταση όπου όλα θα κατευθύνονται τελικά από ε, εταιρείε τη αλλοδαπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώ επειδή θα αφήσουμε τα πάντα να λαμβάνουν χώρα μόνο του στην αγορά. Ναι, θα ήταν πολύ θετικό το να μπορούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουμε ένα εναρμονισμένο μοντέλο όπως αυτό εναρμονίζουν, ε, ε, εφαρμόζουν συγγνώμη, οι Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, και αυτό αποτελεί και μια σημαντική διάσταση της όλης συζήτηση, στην οποία δεν αναφέρθηκα εγώ σήμερα εδώ το απόγευμα. Δηλαδή, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, ο οποίος εξελίσσεται με πολύ αργούς ρυθμούς, γιατί βέβαια θα χρειαζόταν και μια κοινή διαχείριση εναέρης κυκλοφορία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλαμε να ε, κινηθούμε προ τα εκεί. Και αυτό βέβαια τελικά θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αν θα υπάρξει δηλαδή στρατηγική ή όχι. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν εκείνα σε κάποια φάση, αν τελικά επιθυμούν να υπάρξει περισσότερη εναρμόνιση, ενοποίηση, για παράδειγμα, των, ε, ε τη νομοθεσίας τη φορολογικής, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και ούτω εάν επιθυμείτε μια πιο ολιστική προσέγγιση, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι από τα όσα μας είπατε, τότε ε, θα πρέπει να υιοθετηθεί προτού ανοίξει περισσότερο η αγορά των αερομεταφορών προς τα έξω. Μία σύντομη ερώτηση. Αυτή ήταν και η δική μου, οπότε με συγχωρείτε, αλλά ήθελα όχι για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, αλλά για να πάω ένα βήμα παρακάτω ποια θα ήταν η ιδανική κατάσταση, ποιο θα ήταν το ισότιμο παιχνίδι σε ένα κλάδο. για τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αν μιλάμε για ισότιμους κανόνες παιχνιδιού στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιστεύω πως πολλά έχουν ήδη εναρμονιστεί για τον κλάδο. Ως βασική υπηρεσία μέσω αυτού του κανονισμού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο. Περαιτέρω εναρμόνιση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει εναρμόνιση των άλλων τμήματων που επηρεάζουν το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν το ανέφερα, παρόλο που είναι σημαντικό. Και βρίσκεται στα σχόλια που κάνατε για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περιβάλλον. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι που θα προστατεύει και το περιβάλλον που επηρεάζεται από τις ε, εκπομπές, από το θόρυβο κτλ. Αυτά. Ωραία λοιπόν. Και εγώ μία παρατήρηση να κάνω μόνο για τους ισότιμους κανόνες παιχνιδιού με το εργασιακό και το φρολογικό και το περιβαλλοντολογικό δίκαιο είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να προσθέσω εδώ πως τις προτινόμενες ε, τροπολογίες του κανονισμού αυτού που μιλά για το διεθνή ανταγωνισμό έχουμε θέματα εργασιακά, περιβαντολογικά, τα οποία προσπαθούμε να τα εισάγουμε στο κείμενο και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι λανθασμένο. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ε, τόσοι πολλοί κλάδοι που δεν χρειάζονται να είναι οι ίδιες οι συνθήκες εργασιακές παντού. Οπότε εδώ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο και για το διεθνώς περιβάλλον προσπαθούμε να τα δούμε μέσω των, ε, του European Trading System Γίνεται κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο ΙΚΑΟ, αλλά δεν θα έπρεπε να μπουν εδώ σε αυτόν τον κανονισμό. Νομίζω είναι λάθος τόπος. Πολύ ωραία. Τους είχαμε καλέσει. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν. Θα μας είχαν πει και αυτοί οι δύο λόγια. Σας ευχαριστώ. Εάν Θέλεις να... Θέλετε μπορείτε να μείνετε να ακούσετε και τα επόμενα που θα πούμε. Ελπίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν στενοχωρήθηκε που δεν θα σε έκανε κανείς ερωτήσεις, αλλά τώρα έχετε αναλάβει εσείς τα ενία για τα επόμενα. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς της υπηρεσίας μας. Σας ευχαριστώ για την προετοιμασία που κάνατε. θα σας παρουσιάσουμε όταν έχουν κλείσει και τα έγγραφα. Είναι έτοιμοι, περνάμε στο 22. Διατήρηση του ανταγωνισμού στο χώρο των εναριών μεταφορών και ο κύριος Τρεμόσα είναι ο συγητής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντα ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα το γεγονό ότι διοργανώσαμε αυτό το εργαστήριο ακριβώ πριν από τη συζήτηση αυτού του σημείου, γιατί οι παρουσιάσει που ακούσαμε ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσε και ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τη σημασία του ζητήματο το οποίο συζητάμε. Με αυτές τις 42 ε, ε, τροπολογίες που λάβαμε για αυτή την έκθεση και οι οποίες ε, βελτιώνουν ουσιαστικά το κείμενο, ουσιαστικά θα έχουμε μια πολύ καλύτερη τελική γνωμοδότηση από την πλευρά του κυρίου ε, Πίπερ. Όπω είχα αναφέρει εγώ και τον περσινό Δεκέμβριο, εμεί υποστηρίζουμε στεναρά την πρόταση ε, τη Επιτροπή για αναθεώρηση του κανονισμού 868. Με τι λόγω τροπολογίε, λοιπόν, θεωρούμε πω βελτιώνουμε αυτή την πρόταση και καθιστούμε τι σχετικέ διαδικασίε έρευνα και προσφυγή ευκολότερε, όταν δηλαδή υπάρχουν αθέμητε ε, πρακτικέ από την ε, επιχειρήσεων. Ε, και δεν μπορούμε βέβαια να την θεωρήσουμε ως απλώς και μόνο προστατευτική, δηλαδή ως μια πρόταση η οποία προωθείται προστατευτισμό. Και εγώ το λέω σε φιλελεύθερος αυτό. Ουσιαστικά η ε, αερομεταφορές τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει απλώ να προστατεύονται, θα πρέπει πραγματικά να συνεχίσουν να εξελίσσονται αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, και γι' αυτό βέβαια ζητώ να ισχύουν ίσοι όροι του παιχνιδιού στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια αγορά αερομεταφορών και γι' αυτό αξιώνουμε την διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των αερομεταφορών όταν λαμβάνουν κρατικέ ενισχύσει. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι μεταφορεί στην δικιά μα τεράστια αγορά των 500 εκατομμυρίων επιβατών και κατά συνέπεια θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι ο ανταγωνισμό στην αγορά μα λαμβάνει χώρα επί ίση όρη. Όταν κάνουμε λόγο ή όταν κάνω εγώ λόγο στα στην δική μας αγορά. Αναφέρομαι ακριβώς στο γεγονός ότι προσελκύουμε τους ξένους αερομεταφορές επειδή έχουμε όλη αυτή την τεράστια αγορά των ειδικών ε, επιβατών, 500 ε, εκατομμυρίων και με αυτόν τον τρόπο ε, εάν λάβουμε υπόψη μας και την αύξηση της, της, των αερομεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα όσα ε, συζητούνται αυτή την περίοδο στο πλαίσιο των συμφωνιών ε, της Εμπορικής Ένωσης. Κατά δική μου άποψη χρειάζεται ε, οπωσδήποτε η σχετική διαφάνεια έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να ανταποκριθεί ε, στι αρμοδιότητε σε ό,τι αφορά δηλαδή διαφάνεια πάντοτε σε σχέση με αυτές τι κρατικέ ενισχύσει. Επίση, θεωρούμε ότι οι αερομεταφορείς ε, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν κατά της επιτροπή, εάν εκείνη αποφασίσει να τους να ανακαλέσει την άδεια του με βάση μια ε, διαδικασία έρευνα. Ε, και επίση ε, προτείνουμε οι σχετικέ έρευνε να γίνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα, όχι σε δύο αλλά σε ένα έτο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας και τις οποίες θα διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών προκειμένου να τι συμπεριλάβει στη δική του νομοδότηση. Ευχαριστώ. Κάθε πράγμα στον καιρό του, για να το πω έτσι. Καταρχήν να δώσουμε το λόγο στους εστιώδεις ηγητές, ε, ο λόγος λοιπόν στους συνάδελφους Δερουλούν και μετά στους πολύπους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ ε, και εμείς ε, θέλουμε να στεφτεί με επιτυχία αυτή έκθεση του Ραμών. Πάντοτε θέλω να είμαι παρόν όταν παίρνω το λόγο ο Ραμών. Πρόκειται λοιπόν τώρα για μια τεχνική έκθεση, οπότε εμεί υποβάλλουμε μόνο τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίε δύο και βέβαια εδώ βασιζόμαστε στα όσα ήδη γνωρίζει και στην στην κρισία του συντάκτης ε, γνωμοδότησης, ε, εκείνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να εξορροπήσουμε, αν θέλετε, τις ε, πτυχές που καλύπτει επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπή. Είναι τα με τα όσα εμεί θέλουμε να πούμε, αλλά πραγματικά εμπιστεύουμε πλήρω τον αραμών ω συντάκτη γνωμοδότησης προκειμένου να στεφτούμε με επιτυχία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω. Πρόεδρο, δεν υπάρχει άλλο θητή που να θέλει να πάρει το λόγο, οπότε ο Wolfgang που παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ραμόν για αυτή την έκθεση. Ουσιαστικά δεν έχω πολλά σχόλια, δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Ε, καταρχήν σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει να απομακρυνθεί από ορισμένα υποστηρικτικά μέτρα επειδή θα θεωρήσει πως κάτι τέτοιο, επειδή θεωρεί πως κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω σε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή να είναι υποχρεωμένη να έρχεται σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και από εκεί και μετά να λαμβάνει τη σχετική απόφαση. Προφανώ η αρμοδιότητα για τη λήψη τη σχετική απόφαση ε, θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να έχει το δικαίωμα μια διαβούλευση ε, ε, το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, λέω πρώτο. Συνεχίζω και εγώ στα γερμανικά. Η Επιτροπή θέλει μήπω το λόγο. Yeah, the Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. με κυρίες και κύριοι, κύριε Σιγητά, ευχαριστώ πολύ για το σοφές μήνυμα που στέλνετε προς την ε, Επιτροπή Μεταφορών και βεβαίως με μεγάλη προσοχή θα εξετάσουμε αυτές τις τροπολογίες. Άρα, να το εγκρίνουμε ήδη. Διαβόης. Θες να πεις κάτι, Ραμόν. <laughs> αρκεί, αρκεί. Das ist Ε, δεν έξω θα τελειώναμε τόσο γρήγορα. Η δεν θα είχα πιέσει να τελειώσει πιο γρήγορα η ομάδα εργασία για τον ανταγωνισμό. Βλέπετε, καμιά φορά είναι πολύ αποτελεσματική η συνεργασία. Ε, μπορεί να έχουμε και κάποιε μεγάλε διαφωνίες και καυγάδες άμα παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας θα έχετε την ευκαιρία να τα απολαύσετε όλα αύριο το πρωί λοιπόν έχουμε την οδηγία υπηρεσιών πληρωμών που έχει προξενήσει αρκετό άλλο μέχρι